Καλημέρα συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην τελευταία συνεδρίαση πριν από τις διακοπές. Έχουμε λίγη δουλίτσα ακόμα. Ξεκινήσουν οι διακοπές. Υπάρχει καμία παρατήρηση για την ημερήσια διάταξη. Μάλλον όχι. Οπότε... Στο σημείο 21 το θέμα περί Πολωνίας νομίζω μπορεί να μη συζητηθεί γιατί το έχουμε συζητήσει ήδη τον Ιούνιο. Κατόπιν Είμαστε, ξέρετε, και Επιτροπή Υγείας. Και σήμερα υπάρχει αιμοδοσία του Ερυθρού Σταυρού στο Κοινοβούλιο και οι συνεργάτες μας. Καλά, μπορεί να δώσει και κανένα βουλευτή άμα θέλει αίμα. Γιατί όπως ξέρετε πάντα υπάρχουν λήψει στο αίμα. Δεύτερον, μπορώ να σας πω τι έγινε στη, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών ε, Περιβάλλοντος χτες και προχτές στην ε, Πολωνία. Πρώτο θέμα αποτελεσματική χρήση πόρων. Εκεί πέρα η Κομισιόν αρχές Σεπτεμβρίου θα υποβάλει έναν οδικό χάρτη και θα, κάνουμε, θα υποβάλουμε και μια έκθεση προσεχώς. Δεύτερο θέμα έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δράσης. Υπήρχε πολλή συζήτηση για το τι θα πρέπει να περιέχει, αλλά τελικά επιθυμία όλων ήταν να υπάρξει έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Τρίτο θέμα ήταν η προστασία του κλίματος και η προετοιμασία για τον Τέρμπαν. Εδώ πέρα τονίστηκε πως ε, πρέπει να θεωρηθεί και ως μια αφρικανική διάσκεψη και να συζητηθούν ζητήματα όπως η ενεργειακή πολιτική, η ΑΠΕ όσον αφορά την Αφρική, προστασία των δασών. Ε, συμφωνία δεν θα υπάρξει ούτε στον Τέρμπαν γιατί ο Ομπάμα ξεκαθάρισε πως ε, πριν τις προεδρικές εκλογές δεν θα κάνουν τίποτα ε, οι Αμερικανοί, οπότε ούτε στο Ντέρμπαν θα έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία. Äh, äh, Επίσης αναφέρθηκε η έκπληξη και η απογοήτευση για το ότι το Κοινοβούλιο δεν πέρασε το ψήφισμά του γιατί απ' έξω αυτό θεωρείται ως μη ενότητα στον τομέα της ε, προστασίας του κλίματος και πράγματι βεβαίως είναι αξιοσημείωτο ότι στην Επιτροπή μας ε, έχουμε συμβιβασμό όλων των ομάδων και η οποία μετά δεν στέκει στην Ολομέλεια και πάνε μέλη της Επιτροπής μας και καταθέτουν τροπολογίες κατά του συμβιβασμού αυτού. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε γιατί η έκθεση Eichhout, ε, στην έκθεση Eichhout αφιερώθηκε πολλής χρόνος, ενέργεια, δουλειά. Μία φορά ήδη απέτυχε στην Ολομέλεια, για... έχουμε ήδη αποτύχει για την ασφάλεια δηλαδή των πυρηνικών σχεδίων. Τώρα για την συνέχεια της προστασίας του κλίματος ε, δεν γίνεται να γίνεται συνέχεια αυτή η δουλειά. Ε, πρέπει νομίζω να το συζητήσουμε αυτό. Δεν ξέρω. Να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, ένα σχέδιο Β. Δεν είναι δυνατόν να καταστρέφονται αυτές οι θέσεις και η δουλειά που έχει γίνει και νομίζω πως βγήκαμε εξασθενημένοι και όχι ενισχυμένοι από αυτή την υπόθεση. Θέλει κάποιο τον λόγο επ' αυτού, ο Ρίχαρτ Ζέμπερ και μετά Νταν Γιώργενσεν. Ναι, καλημέρα. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη τώρα να συζητήσουμε μια έκθεση η οποία έχει ήδη ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Αυτό ήθελα να πω. Α, τώρα για την ομάδα μου να πω ξεκάθαρα πως εμείς στηρίσαμε τον συμβιβασμό που επετεύχθη. Ήταν σαφές πως το έχουμε τονίσει και πολλές φορές πως ε, για εμάς ε, το 20% είναι μείωση είναι ένα 5% από ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Τώρα αν έρχονται ενοποιημένες τροπολογίες που γράφουν 30% ήταν σαφές ε, πως ε, θα ψηφίζαμε κατά. Είχαμε ψηφίσει κατά και στην Επιτροπή. Η αξιολόγηση της ε, ψηφοφορίας δείχνει πως ε, έγινε δεκτή η έκθεση από τα περισσότερα δικά μας μέλη, αλλά από άλλες ομάδες μετά από δύο πλευρές ε, ε, υπήρχε μία επίθεση ε, γιατί εντάξει κάποιοι θεωρούσαν δεν πήγε αρκετά μακριά, για κάποιους πήγε πάρα πολύ μακριά. Οπότε ήταν νομίζω σαφής, διάφανη η θέση του Έλκεσας. σας υπήρχε και στη διάθεσή σας ένας κατάλογος με τις κόκκινες γραμμές της δικές μας, οπότε δεν υπήρχε καμία έκπληξη. Οπότε το μήνυμα το οποίο έστειλε το Κοινοβούλιο δεν νομίζω να είναι κάποια εξασθένηση, αλλά ξεκάθαρα εξέφρασε ε, την άποψη του Κοινοβουλίου πως 30% θα πρέπει να έρθει μόνο όταν έχουμε μια διεθνή συμφωνία. Αυτή ήταν πάντα η γραμμή μας. Γι' αυτό, όπως είπα, εμείς θεωρούμε πως ε, έχουμε ενισχυθεί και όχι εξασθενήσει και ελπίζω αυτή η ερμηνεία ε, να είναι και η ερμηνεία του Πρόεδρου για τα γεγονότα. Κοιτάξτε, ναι, ε, θα μιλήσει τώρα ένας από κάθε ομάδα. Ε, δεν είχαμε προβλέψει πράγματι συζήτηση. Ήταν Γιώργενσον. Εκπλήσω με λίγο που ακούω το Ζέμπερ να λέει πω η γραμμή τη ομάδα του ήταν διάφανη. Γιατί προφανώς δεν ήταν. Για μας είχαμε ένα συμβιβασμό για, για τους άλλους δηλαδή. Είμαι ευρωβουλευτή τώρα εδώ και 7 χρόνια και σκιώδης εισηγητής σε πολλές εκθέσεις και ποτέ δεν έχω δει συμβιβασμό όπου μετά μία από τις μεγαλύτερες ομάδες δεν, δεν τον υπερασπίζεται στην Ολομέλεια. Εντάξει, μπορεί να έχει συμβεί καμιά φορά, εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε συμβιβασμό για το 25% εσωτερικό. Ήταν επίσης σαφής η αντίληψη όλων των ομάδων πως πέρα από αυτό το συμβιβασμό θα υπήρχε μια ενοποιημένη τροπολογία Τη οποία δεν αποτελούσε μέρο το ΕΛΚ, αλλά ο εισηγητή του ΕΛΚ το ήξερε και το είχε αποδεχτεί. Και δεν είχε πει πως μετά αυτό σημαίνει πως δεν θα στηρίζονταν πλήρως η τροπολογία. Το είχε πει ρητός αυτό στις διαπραγματεύσεις. Εντάξει να μην συμφωνούμε να μην μπορούμε να φτάσουμε σε συμβασμό, αλλά δεν είναι σωστό να λέμε πως έχουμε συμβασμό και μετά να πάμε στην Ολομέλεια και ξαφνικά να μην ε, υπάρχει συμβασμός. Και βεβαίως γι' αυτό καταψηφίστηκε ε, η έκθεση. Προφανώς πρέπει να καταψηφίσουμε μια έκθεση εάν ο συμβιβασμός στον οποίο βασίζεται ολόκληρη η έκθεση δεν, περνάει. Ναι, Μπάς Άικχαουτ. Δεν θέλω το. Θέλω να ανοίξω τη συζήτηση γιατί ψηφίσαμε. Έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση τώρα. Αλλά θέλω τελικά να τα καταγράψουμε σωστά τα πράγματα στην Επιτροπή Ένβη και σε όλες τις ε, συναντήσεις. Ε, πριν από αυτό είχαμε ανοιχτή συζήτηση με τους σκιώδεις και είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Και συμφωνήσαμε σε ένα σημείο να διαφωνήσουμε. Και αυτό ήταν στις 30. Και προηγουμένως εσωτερικά ήταν το 30%. Και συμφωνήσαμε ε, να ε, με το ECR και το ELK σε αυτή την τροπολογία. Έτσι λοιπόν το 30% εγκρίθηκε και ξέραμε ότι είναι μια ενοποιημένη τροπολογία, δεν ε, εγκρίθηκε από όλους λοιπόν και ξέραμε ότι θα ήταν στενή η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ψηφορία στην ΕΝΒΗ υπήρχαν και πάλι τροπολογίες που κατατέθηκαν και ξανά άνοιγαν ε, και πάλι τους συμβεσμούς και εγώ είπα ότι αυτό είναι επικίνδυνο γιατί και πάλι ξανανοίγουμε κάποιου συμβασμού του οποίου είχαμε καταλήξει πριν. Και αυτό ήταν πάρα πολύ διαφανέ και συμφωνώ με τον Ρίτσαρτ ότι ήταν διαφανέ. Ξέρω ότι ήταν και τροπολογίε, αλλά και εγώ πολύ ανοιχτά είπα ότι δεν μπορούν να εγκριθούν αυτέ οι τροπολογίε από του υπολείπου, από άλλου. Έτσι λοιπόν, υπήρχε ένα στίχημα σκόπιμο να υποστηριχτεί αυτή η έκθεση από αυτή την τροπολογία, η οποία πράγματι άλλαζε το συμβασμό επί το οποίο είχαμε συμφωνήσει προηγουμένω. Αυτό για τα πρακτικά. Και να πω ότι είχαμε πάρα πολύ καλέ διαπραγματεύσει, ήταν όλε διαφανεί και σε κάποιο σημείο συμφωνήσαμε να διαφωνήσουμε. Και αυτή θα έπρεπε να είναι ψηφοφορία στην Ολομέλεια και είναι κρίμα που κάποιε από τι τροπολογίε επανέρχονται τώρα για το συμβασμό επί το οποίο συμφωνήσαμε και κατά τη διάρκεια των μετά Ευχαριστώ. Ναι. Ε, ας μιλήσει ένα από κάθε ομάδα και ο Μύρο Λαβούτσκι για να μην... Ε, τώρα, ναι, εντάξει, να μην γίνει συζήτηση, αλλά κάντε δηλώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μα δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Θόρυβος επικρατεί. Λοιπόν, να πω λίγα λόγια για το ECR. Πρέπει να τονίσω πως οι διαπραγματεύσεις για αυτή την έκθεση ήταν φιλικές και ειλικρινείς, αλλά πρέπει να τονίσω πως από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει πως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε πρόταση που πάει παραπέρα από την πρόταση της ε, Κομισιόν. Και μάλλον ε, ο συμβιβασμός θα ήταν γύρω στο 25, παρά το ότι η δική μας θέση ήταν η αρχική θέση της Επιτροπής 20-20-20, εάν δεν υπάρξει παγκόσμια συμφωνία. Δεν έχει επιτευχθεί αυτή, οπότε λέμε εντάξει, αν είναι στο πνεύμα του συμβιβασμού του Κοινοβουλίου να πάμε στο 25, αλλά όχι παραπέρα. Οπότε νομίζω πως θα συμφωνήσει και ο εισηγητής πως ε, αυτή η θέση τονίστηκε σαφώς ε, ε, στην συνάντηση των σχεδόν εισηγητών από την αρχή και δεν ε, συμφωνώ ε, όταν υπάρχει μια έκθεση που δεν έχει εγκριθεί ότι είναι πρόβλημα, ε, αυτό είναι μέρος της δημοκρατίας. Και ένα ήταν το μήνυμα, πως η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν θα συμφωνήσει να πάει παραπέρα. Και δεν νομίζω να είναι πρόβλημα αυτό και το τι εντύπωση δίνουμε στους υπουργούς περιβάλλοντος, αυτή είναι η δημοκρατία. Μάλιστα. Όπως σας είπα, εγώ το θεώρησαν αδυναμία του Κοινοβουλίου και το θέμα δεν ήταν το 30%, ήταν το τι περιέχεται στο νοδικό χάρτη του 2005 της ε, Κομισιόν για το κλιματικό πακέτο του 2008 που σημαίνει 50% εσωτερική μείωση. Αυτό ήταν στον συμβασμό, δεν πέρασε στην Ολομέλεια. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Ε, η κυρία Γιώργαν Σίσελη ήταν σκιώδης εισηγήτρια. Τέλος μίλησε κάθε ομάδα, αλλά είναι και η Επιτροπή Βιομηχανίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω και εγώ ως εισηγήτρια στην Επιτροπή ΤΡΕΠ. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η εκθέση αυτή προετοιμάστηκε με το άρθρο 50 και αυτό σημαίνει οι μικτές αρμοδιότητες ε, είναι και και αυτό σημαίνει ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την έκθεση, όχι μόνο από την Επιτροπή ΕΝΒΗ, αλλά και από την Επιτροπή ΤΡΑ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Άικουτ. Ήταν διαφανής και ανοιχτή διαδικασία, αλλά η τελική απόφαση της ΕΝΒΗ δεν ήταν ένα συμβασμός μεταξύ ΤΡΑ και ΕΝΒΗ. Και ε, πιθανότατα αυτό είναι και ένα από του λόγου. για αυτή την κατάληξη. Έτσι λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρότεινα να αλλάξει και η πολιτική μας τάση, να προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε και ένα συμβιβασμό και συμβιβασμό με την Επιτροπή με την οποία έχουμε μικρές αρμοδιότητες. Δηλαδή υπάρχει και στο ιστορικό της έκθεσης μια τέτοια γραμμή. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε φιλικοί άνθρωποι, ας μιλήσει ο Καλχάιτς Φλόρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσει να, να ακούγεται πως δεν τηρήθηκαν οι συμβιβασμοί. Εγώ και στην Επιτροπή καταψήφισα το 25% γιατί όλοι αυτοί οι όροι, όλο αυτό το νόημα του, του 25% για εμένα ήταν πολύ ομιχλώδες. Δυστυχώς το έλαβα μόνο στα αγγλικά, γι' αυτό καταψήφισα και στην Επιτροπή αγαπητέ φίλε και πρόεδρε που με κατηγορείτε. Εγώ καταψήφισα και στην Επιτροπή. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ε, όσον αφορά και τον πρόεδρο. Ε, λυπούμε που έζησε κάτι τέτοιο ο συνάδελφος ο κύριος Άικχαουτ, γιατί εργάστηκε καλά, δεν, δεν ζήτημα. Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε λίγα σημεία, αλλά κύριε πρόεδρε, γιατί γράψαμε τελικά αυτή την έκθεση. Δηλαδή, επιστρέψαμε από την Κανκούν και θέλαμε να περάσουμε το 30% παρά το ότι δεν το συζητήσαμε καν στην Κανκούν. Δεν ήταν θέμα συζήτησης στην Κανκούν. Κύριε Πρόεδρε, ακόμη λιγότερο θα αποτελέσει θέμα διαπραγμάτευσης στον Τέρμπαν. Θα είναι όλα ή τίποτα, όχι το 30%. Εάν δεν έχουμε εκεί πέρα συνθήκη, την οποία ήδη είπατε ότι δεν θα έχουμε λόγο των Αμερικανών, θα είναι καταστροφική η κατάσταση. Χρειάζεται ένα μέσο μετά το, το Ντέρμπαν. Εντάξει δεν επιτρέπεται πλέον να λέγεται Κιώτο γιατί έχει καεί η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει το Ντέρμπαν δεν είναι πια, στο Ντέρμπαν δεν είναι πια το ζήτημα το 30%. Το θέμα είναι αν θα ε, καταρρεύσει το έργο 20 ετών ή αν θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Είναι τελείως διαφορετικά τα ζητήματα που παίζουν εκεί πέρα ρόλο. Γελάνε μαζί μας οι Αμερικάνοι όταν λέμε πώς θα πάμε στο 30% εθελοντικά. Λένε, μου λένε μα πού τα βρίσκεται αυτά τα πράγματα, κάνε και 40%. Τι, τι μας ενδιαφέρει εμάς, ούτε και τους Κινέζους ενδιαφέρει. Η απόφαση δηλαδή για να γίνει αυτή η έκθεση δεν ήταν ίσως η εξυπνότερη. Εντάξει. Ε, τώρα αν λέτε πως ε, το έγραψε για τον Τέρμπανο την έκθεση ο Μπασακχάουτ δεν το καταλαβαίνω. Μα αγαπητέ κύριε Καλφρόντς, πραγματικά εσείς είπατε ότι δεν ήταν για τον Τέρμπαν η έκθεση. Όταν πάμε στον Τέρμπαν θα γράψουμε μια έκθεση γι' αυτό. Ήταν αντίδραση στην εσωτερική πολιτική της Ένωσης που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Μια έκθεση η οποία αντανακλά την ανακοίνωση της Κομισιόν ε, τις αναλύσεις και τις μελέτες που έχουν γίνει για το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020 και θέλαμε να τοποθετηθούμε για να ενθαρρύνουμε το ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι θεωρούσαμε ότι θα είμαστε το 2008. Ε, κατέρευσε αυτό και αυτό άρα είναι κατά την άποψή μου μια αποδυνάμωση όταν α, καταρρύπτεται μια τέτοια έκθεση στην Ολομέλεια και δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον θέση του Κοινοβουλίου έναντι του Συμβουλίου. Είδα στην Πολωνία τι τρέχει μες στο Συμβούλιο. Υπάρχουν πολύ φιλόδοξες χώρες και υπάρχουν κάποιες που είναι πολύ πίσω και το Κοινοβούλιο είναι η κινητήριος δύναμη και θα ήταν καλό αυτό το ψήφισμα για ολόκληρη αυτή την ε, αλλαγή. Τόσο χρήσιμο ήταν να μιλήσουμε γιατί είχαμε κάνει τόσο πολύ ε, δουλειά και κατέληξε στον κάδο της ανακύκλωσης. Θα το δούμε τώρα στο επόμενο ψήφισμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξη, σημείο 3. Ε, τα πρακτικά 16 ε, και 7 Μαρτίου, 11 και 12 Απριλίου και 21 Ιουνίου. Εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση εγκρίνονται και περνάμε στις ψηφοφορίες. Ε, Όχι, δεν πάμε στις ψηφοφορίες. Πάμε στις ανακοινώσεις κοινών θέσεων. Το ένα αφορά τα βιοκτώνα, έκθεση κλάς. Έχουμε σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση που θα κατατεθεί 8 Ιουλίου. Έγινε αυτό. Εξέταση σχεδίου συστάσεως για 8 Σεπτεμβρίου, στη δεύτερη ανάγνωση. Προθεσμία 12 ε, Σεπτεμβρίου για τροπολογίες. 4 Οκτωβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή. Και το Συμβούλιο θα καταλήξει σε κοινή θέση 26 με 29 Σεπτεμβρίου και θα μας την μεταδώσει. Μετά έχουμε την έκθεση Florence για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Το ίδιο ακριβώς χρονοδιάγραμμα. Οπότε όπως σας είπα ε, εξέταση θα έχουμε τον τροπολογιών 12 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου μετά θα έχουμε την ε, ψηφοφορία. Μετά, σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι φάσεων εκπομπών ε, στε, στενά, σε ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο. Ο εισηγητή είναι ο Ταταρέλα και έχουμε μια τροπολογία 3, Παύλ Πότς που είναι γλωσσική, τροπολογία 4 και 5 είναι οι ίδιες. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 με προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την αρχική λοιπόν εκδοχή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελκ. Α, δεν είναι σαφές. Μιλάμε για την αρχική έκδοση εκτιμώντας 4α νέο. Κατέπεσε η τροπολογία και τώρα περνάμε στην αρχική εκδοχή 4α νέο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μετά τροπολογία 1. Κατά πίπτη. 7 και 8 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 9 και 10 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Τροπολογία 11 και 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Τροπολογία 2 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρα της ε, ψηφοφορίας 48 υπέρ 5 κατά καμία αποχή Οπότε εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια στον κύριο Ταταρέλα. Πρέπει τώρα να ψηφίσουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Όχι, το είναι ένας παραπάνω από τους φιλελεύθερους. Τώρα είναι εντάξει. 55 υπέρ. Κανείς κατά, καμία αποχή. Τώρα μπορώ να συγχαρώ. Ωραία. Ήταν πολλή δουλειά που έχει γίνει. Και οι ελκυστήρες αυτοί θα χαρούν για το ότι θα έχουν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Περνάμε στο σημείο 7. Έκθεση της Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη για προστασία από τις καταστροφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επίσης τον κατάλογο των ψηφοφοριών και πολλές συμβαστικές τροπολογίες. Πράγμα καλό. Περνάμε συμβαστική υπαριθμόν 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. Ενοποιημένη τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ενοποιημένη 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά περνάμε στις παραγράφους 35 και 36 είναι ταυτόσιμες και συμβατές αλλά πρέπει να τις ψηφίσουμε και τις δύο πρώτα απ' όλα 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά περνάμε στην 38 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή Ρέγγι 1 υπέρ κατά εποχές δεκτή. Δεύε 4 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή επίσης. Αφέτ 5 δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά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 Aber haben wir doch. Πρέπει να ψηφίσουμε την 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Α, καταπίπτει. Μάλιστα. 49 υπέρ. Κατά. Εποχές. Δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 της αφέτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ρέγγι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ρέγγι 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15 τη Ρέγγι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε πέρας 29 με 29 ψήφους δεκτή. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 της ΔΕΒΕ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέγγι 2 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή Ρέγγι 4 με χωριστή ψηφοφορία, μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Ποιος ψήφισε από το ΕΛΚ. Δεν είδα τίποτα. Υπέρ. Πώς... Κοιτάω την εισηγήτρια. Άρα εντάξει έχει γίνει δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ. Της Ρέγγι 4. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 68. Πέρας. Α, είναι σαφές. Δεκτή. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά συνεχίζουμε με την 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 της αφέτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 της αφέτ υπέρ κατά αποχές δεκτή DV5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 84 τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 χωρίς τη ψηφοφορία μέρος πρώτο α ένα μέρος υπέρ του πρώτου μέρους κατά αποχές δεκτό δεύτερο υπέρ κατά Το δεύτερο μέρος καταπίπτει. Οπότε έχουμε πάει στην εννέα της Ντέβε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μετά. Τροπολογία. 12 της Ρέγγι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 92 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές 99 υπέρ κατά αποχές αυτή, 100 υπέρ κατά αποχές αυτή, Ρέγγι 14 υπέρ κατά αποχές αυτή, Ρέγγι 16 υπέρ κατά αποχές αυτή, εκτιμώντας 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή Τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή τέσσερα μπεφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή Τώρα περνάμε στα εκτιμώντα, Ναι, το όχι, την 6 έχουμε ακόμα υπέρ. Κατά. Να αποχές δεχθεί. Οπότε τώρα περνάμε στα εκτιμώντα 7 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Με προφορική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 πίπτη 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή κατόπιν εκτιμώντας δέλτα, το αρχικό με χωριστή ψηφοφορία, πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά εκτιμώντας F χωριστή ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο ποιος είναι υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Καλή ιδέα. Πέρας. Δεκτή. Είκοσι πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ο συνάδελφος Σόνικ παλεύει εκεί με την κάρτα. Ε, κάπου πρέπει να, να λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Τώρα. Όλα εντάξει. Ωραία. Οπότε έχουμε φτάσει στην 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές Οπότε ε, πήγαμε πολύ γρήγορα στην 23 και στην 24 γιατί αναφέρεται πως καταπίπτει αν απορριφθεί το αρχικό κείμενο και αυτό είχε γίνει δεκτό οπότε πρέπει να ξαναδούμε τι γίνεται με τις τροπολογίες ε, Bruyne και Gardini. Οπότε ψηφίζουμε τώρα την 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αυτά λοιπόν. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας με μεγάλη ενότητα 55 υπέρ κανένας κατά καμία αποχή συγχαίρουμε την κυρία Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη είμαστε αρμόδιοι και για την προστασία από καταστροφές ε, κάτι το οποίο είναι τόσο ορατό εδώ στην Επιτροπή μας αλλά είναι μια μεγάλη έκθεση για την καλύτερη προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, από τις ε, καταστροφές στις γειτονικέ φορές και παντού στον κόσμο. Περνάμε τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού ένα νέο μέσο όπου δικαίως ως Επιτροπή ε, φραστήκαμε κι εμείς γιατί ο οικονομικός συντονισμός ε, και η φορολογία θα πρέπει να λάβει υπόψη πτυχές της αηφορίες ε, και να παίξει ρόλο σε όλα αυτά. Ο Κρεσέντσο Ριβελίνη είναι συγητή. Έχουμε τον κατάλογο των ψηφοφοριών τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεκτή. Ε, να το ξαναδούμε. Πέρας. Δεκτή, ναι. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4 και 5 ταυτόσιμες με χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται μάλιστα. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 17 υπέρ. τα αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μικρή διαφορά. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Να αν το θέλετε. 16 πέρας της ψηφοφορίας Ναι, έχετε γερό σήμερα Μετά 9 και 10 ταυτόσιμες, ποιος είναι υπέρ. 9 και 10. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και γίνεται δεκτή. Τώρα λοιπόν ακολουθεί η 11. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 με προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ της 13 με την προφορική τροπολογία κατά αποχές να επαληθεύσουμε Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Μια στιγμούλα. Έχουμε απορρίψει την προφορική τροπολογία. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ της 3. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ να την επαληθεύσουμε απορρίπτεται 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά 25 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και περνάμε άρα στην τελική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. 52 υπέρ. Μία ψήφος κατά τρεις αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Κρεσέντσιο Ριβελίνη. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Συνεχίζουμε Ένα ωραίο θέμα τώρα οι μέλισσες. Τζούλι Γκέρλινγκ είναι η συγγήτρια. Θέλω να αποσύρω την τροπολογία μου, την 148. 148, η κυρία Σίσελη, μάλιστα. Είναι καλό αυτό για τις μέλισσες. Ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι μέλισσες στη φύση και η μελισσοκομεία. Το επιβεβαιώνει και ο Αλόης Πέτερλε που είναι μελισσοκόμος, ο μόνος μελισσοκόμος εδώ μέσα. Ωραία. Kompromiss Nummer 1. Συμβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ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 Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ενοποιημένη 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συνεχίζουμε με την συμβαστική 2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές ναι, δεν είναι σαφές να επαληθεύσουμε την πέντε. Πέρας. Δεκτή. Δέκα. Υπέρ. Κατά. Για αποχές. Τι. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οπότε την επόμενη πρέπει να την ψηφίσουμε χωριστά. Τροπολογία 25 της εισηγήτριας, μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 23 με προφορική τροπολογία υπέρ καταπίπτει 23 Συνεχίζουμε με την 27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τριάντα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τριάντα ένα. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ 34 τέσσερα, είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, εντάξει πέρας Δεκτή. Σαράντα Κατά. Αποχές δεκτή. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 54 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 52 προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 53 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ναι να επαληθεύσουμε την 56 Πέρας. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτή. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ Οι δύο μεγάλες ομάδες είναι υπέρ. Νομίζω ότι θα να την επαληθεύσουμε την 79. Πέρας. Ε, ναι, με, με συγχωρείτε. 80 υπέρ κατά αποχές 81 υπέρ κατά αποχές 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή συνεχίζουμε με την 92 με προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αντελβό ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται να επαληθεύσουμε Beendet. Πέρας. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. κατά αποχές δεκτή 98 με προφορική τροπολογία χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές να υπαλληθεύσουμε 98 πρώτο μέρος με προφορική τροπολογία. Να πολιτεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε την 115. Ποιος είναι υπέρ. να επαληθεύσουμε. Πέρας. Δεκτή. 122. Νέα προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της 122. Κατά. Αποχές δεκτή. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Δεκτή. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίντα ενοχλεί τώρα αυτό λίγο. Συγγνώμη. Έχει ενοχλεί, ενοχλεί πραγματικά. 74 προφορική τροπολογία καταπίπτει 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 108 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συνεχίζουμε με την 114. Ποιος είναι υπέρ. συζητηθεί. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. οπότε είναι λίγο περίπλοκο. Πρέπει να ψηφίσουμε την 101 από ό,τι μου λένε εδώ πέρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 126 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά αποχές δεκτή 128 υπέρ κατά αποχές δεκτή 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές δεκτή 131 υπέρ κατά αποχές δεκτή 132 υπέρ κατά αποχές δεκτή 140 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 134. πέρας. Δεκτή. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές δεκτή 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή 146 υπέρ κατά αποχές δεκτή 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 48 αποσύρεται, άρα 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 150. Παύλ Πότς. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή και 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η συγκίτρια έχει το λόγο πριν την τελική ψηφοφορία. Έχει τον λόγο. Um, Ευχαριστώ. Βρίσκομαι σε μια συνήθιστη θέση να ψηφίζω κατά της δικής μου γνωμοδότησης και θα το εξηγήσω. Μπορείτε να δείτε πόσο ενδιαφέρον υπήρχε για την έκθεση αυτή και είχαμε συμφωνήσει σε κάποια σημεία, αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω για ένα κείμενο το οποίο λέει ότι γενετικά τροπομένοι οργανισμοί ιδίω πλήντουν ε, τις μέλισσες όταν δεν υπάρχουν ε, τέτοια αποδεικτικά στοιχεία και αυτό υπάρχει σε κάποιες ε, τροπολογίες ε, η διατύπωση ε, τελικά μέσω της διατύπωσης αναφέρονται θέματα για τα οποία δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία και εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρ' όλα αυτά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας 32 υπέρ 17 κατά 7 αποχές Συγχαρητήρια παρόλα αυτά θα χαρούν οι μέλισσες. Σε όλη την Ευρώπη. Και ξέρουν αυτές καλύτερα εάν βλάπτουν οι γενετικά τροπημένοι οργανισμοί ή όχι. Περνάμε τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Εξυγχρονισμός πολιτικής μουσείων συμβάσεων, Άσα Βέσλοντ, έχετε τον κατάλογο των ψηφοφοριών και ξεκινάμε με την συμβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 2 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ενοποιημένη 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ναι, θα το επαληθεύσουμε. Abstimmung beendet. Πέρας και γίνεται δεκτό. Οπότε παραμένει η 10 Κρήτον Αρσένης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. 13 είναι γλωσσική. 17. Α, όχι. Συμβαστική 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεκαεφτά υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή ενοποιημένη 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ενοποιημένη τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 51 με χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το ECR δεν είδα τι ψήφισε οπότε να επαληθεύσουμε την 51 μέρος πρώτο πέρας δεκτή Μέρος δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 52 υπέρ. Καταπίπτει, μου λένε εδώ πέρα. 52 Συνεχίζουμε με τη συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία στην παράγραφο 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη 13 υπέρ 13 κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 Συνεχίζουμε με την 70. 70 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή και 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, 68 είπατε ότι υιοθετήθηκε και ψηφίσετε την 72, αλλά η 72 καταπέπτει αν υιοθετηθεί 68 καθώς πρόκειται για διαγραφή η 68, οπότε δεν έχει νόημα να ψηφίσουμε την 72. Πράγματι, πράγματι, ωραία, δεν ισχύει η ψηφοφορία. Καλά το είδατε. Οπότε, ψηφίσαν όλοι, πέρας, 49 υπέρ καμία εποχή κανένας κατά. Συγχαίρουμε τον Άσο Βέστλοντ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Ξέρετε πως οι συμβάσεις του δημοσίου είναι ένα 25% και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αηφόρο άρα ανάπτυξη. Πριν έρθει ο πρόεδρος του Συμβουλίου και υπουργό Περιβάλλοντος Πολωνίας έχουμε ένα σημαντικό θέμα ακόμα το ψήφισμα. Προφορική τροπολογία για τη μεγάλη διάσκεψη για τη γη που λέγεται Ρίο Θα ψηφίσουμε και θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση ποιος είναι υπέρ. Κατά άποχες ομόφωνα συγχαρητήρια στους ερωτώντες από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και 25 λεπτά συζήτηση τώρα για το ψήφισμα το οποίο υποβλήθηκε. Καρλ Χάιντς Φλόρεντς. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σωστά είπατε, πρόκειται για την σύνοδο της γης. Ε, ξέρετε πως η πρώτη ήταν το 92 στο Ρίο. Εγώ ήμουν τότε φρέσκος ευρωβουλευτής και συμμετείχα και σήμερα πρέπει να πω πως τα όσα έχουν συμβεί στο ενδιάμεσο είναι θλιβερά γιατί δεν έχουμε προχωρήσει πολύ γιατί το ζήτημα της αηφορίας και στις χώρες μας δεν είναι τόσο σημαντικό και σε κάποιες χώρες υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες ε, δραστηριότητες ε, αλλά εντάξει σε περιφερειακό επίπεδο είναι καλά τα πράγματα αλλά δεν υπήρχε καμία μεγάλη επιτυχία οπότε πρέπει να γίνουν καλύτερα τα πράγματα κύριε Πρόεδρε η διάσκεψη αυτή ξέρετε πως ε, μας ενημέρωσε η γραμματεία για το έγγραφο της Κομισιόν την προηγούμενη Τετάρτη και ε, μας είπαν μετά πως θα έπρεπε την Πέμπτη να καταθέσουμε ήδη τις ε, τροπολογίες. Δεν ξέρω, μου θυμίζει κάτι μεγάλες αμερικανικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις που περνάνε τα πάντα βιομηχανικά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να καταθέσουμε τις τροπολογίες. Ε, τουλάχιστον υπήρξε μια αναβολή, αλλά Πρέπει να σκεφτούμε αυτή την πίεση που υφιστάμεθα. Εγώ να μιλήσω με τους υπεύθυνου, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε από την Κομισιόν, όχι μόνο ε, εσωτερικά εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά παρόλα αυτά, Ήδη με πολλούς συναδέλφους ε, γράψαμε νομίζω ένα καλό έγγραφο θέσεων. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο γιατί τώρα οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες που καταθέτουν δεν έχουν και, και πάρα πολύ νόημα. Όλα αυτά, εντάξει, το διαμορφώνω ο καθένας με ανάλογα με το γούστο του. Αλλά ε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι κάποιες βασικές αρχές. Δεν καταφέραμε ποτέ πραγματικά να έχουμε μια συνολική προσέγγιση αηφορίας. Ε, έχουμε δει τους τρεις πυλώνες και τον καθένα χωριστά, αλλά στο μέλλον και τους τρεις πυλώνες, δηλαδή περιβάλλον, κοινωνικά και οικονομία, να τα δούμε από κοινού. Και αυτό οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της συζήτησης νομίζω θα μπορέσουμε να το δούμε καλύτερα. Οπωσδήποτε η βιομηχανία έχει μεγάλη ευθύνη, η οικονομία, γιατί χωρίς πρώτες ύλες δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά και αντιστρόφως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον κόσμο σε όλες τις περιοχές αυτού του πλανήτη. Και όπως σας είπα δεν είναι δυνατόν να συζητιόνται αυτά τα πράγματα στις 12 παρα 5. Εντάξει, έχουμε κάνει όλα μας τα, τα λάθη. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους, σε τελική ανάλυση θέλουμε καλύτερη ζωή και όπως σας είπα για τους ανθρώπους και για το κοινωνική πτυχή και για την οικονομία οπότε πρέπει να ορίσουμε καλύτερα τους στόχους με τους συμμετέχοντες. Γιατί ξέρετε πως ε, συχνά Καμιά φορά είμαστε κατά της, μεγάλη, της μεγάλης του πλήσιμου. Για τα μέσα τώρα μέτρησης, εντάξει, καλό το ΑΕΠ, αλλά δεν περιγράφει τα πάντα. Τα μέσα τα οποία χρειαζόμαστε πρέπει να επεκταθούν, να γίνουν πιο σύγχρονα. Ε, για τη συμπερίληψη των πολιτών, την ανέφερα ήδη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για εφορία, στη συζήτηση αυτή, να δούμε και τις ε, χώρες, π.χ. όταν μιλάμε για εξόριξη μεταλλευμάτων και άνθρακα, να εμπλακούν διάφορες χώρες, γιατί υπάρχουν μεγάλες πολυεθνικές ε, οι οποίες ε, εξορίσουν και δεν δίνουν καμιά σημασία. Δεν μπορούμε να τα αποτεχτούμε αυτό. Πρέπει και οι τοπικές αρχές να συμπεριληφθούν, να έχουν λόγο οι άνθρωποι και οι πολίτες και εν πάση περιπτώσει να κερδίζουν κάτι από όλη αυτή την, την διαδικασία. Ξέρετε, ευχαριστώ να, να μιλάω, αλλά τώρα ευχαριστώ να σας παραδώσω και τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Ναι. Δύο-τρία λεπτά για να μιλήσουμε όλοι. Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, φανταζόμουν ότι θα γινόταν συζήτηση, γιατί έχουμε ψηφίσει, όμως ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία που έχουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε μία απάντηση στο άγγραφο της Κομπισιόν. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο που ουσιαστικά ξαναρχίζει αυτή η συζήτηση γιατί το Ρίο το 1992 ήταν ένα στάδιο πάρα πολύ σημαντικό Είδαμε τι καθορίστηκε λοιπόν τότε και κατόπιν τα επόμενα 20 χρόνια έλαβαν χώρα πολλές εξελίξεις. Έτσι λοιπόν εγώ θεωρώ ότι το έγγραφο της Επιτροπής είναι κάπως ε, περιοριστικό σε σχέση με όλα αυτά που υπάρχουν και σε σχέση με τις προσδοκίες που εγώ νομίζω ότι μπορούν να δημιουργηθούν για το Ρίο 20. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι προέκυψε εδώ. Είδαμε ότι ο πολιτισμός μας δεν είναι βιώσιμος, γιατί βασίζεται σε μια υλική παραγωγή που πρέπει πάντοτε να αναπτύσσεται. Και φυσικά υπάρχουν κάποια όρια στους φυσικούς πόρους και στην ικανότητα της γης να δεχτεί τα δικά μας απόβλητα. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, όχι απλώς να οθήσουμε τον πολιτισμό μας να προχωρήσει προς μια πράσινη οικονομία. Εδώ πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν θέλουμε πράγματι να είναι αηφόρος ο πολιτισμός μας, πρέπει να δράσουμε με πιο ξεκάθαρο τρόπο και να κατανοήσουμε ποια είναι τα θέματα που πρέπει ριζικά να αλλάξουν. Έτσι λοιπόν, ε, όλη τη συζήτηση που ήδη έχουμε ξεκινήσει, εγώ θα την κατευθύνα και πέρα από το ΕΠ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό επιχείρημα για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε αυτή την ε, πλήρη βιωσιμότητα, την καθολική βιωσιμότητα. Έτσι λοιπόν, εγώ επιφυλάσσομαι να παρουσιάσω τροπολογίες γιατί το Ρίο είναι 20 θα είναι ένα ραντεβού πάρα πολύ σημαντικό και εμείς εδώ σε αυτή την επιτροπή είμαστε σε θέση να συνεισφέρουμε ουσιαστικά για την αλλαγή. Ο πολιτισμός μας θα πρέπει να αλλάξει. Αυτός ο πολιτισμός δεν είναι βιώσιμος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λεπάς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι αν επιθυμούμε αυτή η νέα διάσκεψη να είναι συμβολική, να είναι αποτελεσματική. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα που όλοι το θέτουμε, γιατί ε, εδώ και δεκαετίες ε, ουσιαστικά συζητάμε αυτό το θέμα, αλλά δεν συνάδουμε με την πραγματικότητα. Τώρα, το δεύτερο. Η πράσινη οικονομία, ναι, πολύ ωραία όλοι εργαζόμαστε ε, προς αυτή την κατεύθυνση, όμως έχουμε πρόοδο σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη ή την αντικαθιστά κάτι τέτοιο και για τους υπόλοιπους πυλώνες στους οποίους αναφέρθηκε ο συνάδελφος Φλόρενς που βρίσκονται γιατί δεν θα εγκαταλείψουμε τον κοινωνικό και τον περιβολητικό παράγοντα υπέρ της οικονομίας δηλαδή πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πράσινη οικονομία Δεύτερο σχόλιο για τις τεχνολογίες πολύ καλές οι τεχνολογίες, όλοι είμαστε υπέρ, μπορούν να αποτελέσουν ένα τμήμα της λύσης, αλλά πρέπει και να τις αξιολογήσουμε ορθά για να μην έχουμε βραχή κυκλώματα και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θέμα των νανοτεχνολογιών ε, αλλά και στη μηχανική. Φυσικά πολλές ε, μελέτες μπορούν να γίνουν ε, για τα αποτελέσματα, για τις επιπτώσεις και επίσης πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν θα μας λύσει τεχνολογία όλα τα προβλήματα και το τρίτο σημείο θα πρέπει να επεκτείνουμε όλα αυτά στις εργασίες μας σχέση με την ανάπτυξη και το ΑΕΠ. Αν δεν είμαστε ικανοί να τροποποιήσουμε τους δείκτες μας, αν δεν είμαστε ικανοί να βρούμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης βάσει αυτών των δικτών. Φοβάμαι ότι τελικά θα βρισκόμαστε πάντα στο ίδιο σημείο μετά την επόμενη διάσκεψη. Δεν ε, είναι κριτική αυτά που λέω, απλώς ε, αναφέρω την επιθυμία να τα δικαταστήσουμε όλα αυτά σε ένα πιο γενικό πλαίσιο και κυρίως ε, στο πλαίσιο της αποδοτικότητας. Είπαν συνάδελφοι ότι οι γείτονες και φίλοι από την Αμερικανική και την Ασία θα μας κοροϊδεύουν αν ε, παραμείνουμε εκεί. Νομίζω ότι είναι αλήθεια. Θα πρέπει να περάσουμε σε ένα πολύ πιο ενεργό στάδιο σε σχέση με το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπελιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 20 ε, χρόνια μετά ο απολογισμός ε, πονάει. Είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση, είναι ακόμη παρούσα Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ε, ως προς την ανάλυση, αλλά θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας. Σε λιγότερο από ένα χρόνο στο Ρίο θα είμαστε στο ύψος των περιστάσεων, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως κινητήριος δύναμη για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, προκλήσεις που παρουσιάζει η τέταρτη σύνοδος 20 ε, χρόνια μετά το Ρίο και πάνω από 30 χρόνια μετά την πρώτη σύνοδο της γης, ε, τη σύνοδο της Στοχόλμης ή και 40 χρόνια, αν έχω υπολογίσει σωστά. Θα είναι αποφασιστικό στάδιο προς την τον τελικό στόχο. Και στα πλαίσια του σχεδίου, η πράσινη θα ήθελα να καταστήσουμε πιο ισχυρή την πρόταση. Θα καταθέσουμε μέχρι αύριο περίπου 30 τροπολογίες, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα μόνο να πω, γιατί αναφέρθηκε, δεν είναι μόνο καλοπιστική η παρέμβασή μας, θέλουμε να επέμβουμε για θεμελιώδη ζητήματα σε διεθνέ επίπεδο και σε επίπεδο κοινοβουλία έχουμε κάποια κεκτημένα και ίσω πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο ω προς την ε, καινοτομία η σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίση έχει ιδιαίτερη σημασία. Να κατοχυρώσουμε μια νέα αρχή ε, τη μη υποχώρηση ω προ τα περιβαλλοντικά και εκτιμένα, διότι αυτό είναι θεμελιώδες δικαίωμα, να επανέλθουμε στη βιοαιρεσιμότητα των ε, δημοσίων ενισχύσεων και αναθεώρηση των δικτών, δηλαδή του ΑΕΠ, να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μα ω προ την επιστημιστική κυριαρχία, να βασιστούμε συμφωνίες και ίσως ε, να απευθύνουμε έκκληση για νέες διαπραγματεύσεις ε, σε τομείς που δεν έχουν ρυθμιστεί, όπως η ναυτιλία. Και τέλος, όπως και στην Ιαπωνία, χρήσιμο θα ήταν με διπλωματικό τρόπο αλλά με πυγμή να ε, ζητήσουμε από τον αμφιτρίωνα τη Βραζιλία το 2012 στη Σύνοδο του Ρίο να αναλάβει σοβαρή δέσμευση για να σταματήσει η αποψήλωση των δασών στην επικράτειά της. Δεν χρειάζεται, όπως σας είπα, να μπω σε λεπτομέρειες ε, για τις 30 αυτές τις τροπολογίες, οποίες θα καταθέσουμε και που θα συζητήσουμε στη συνέχεια στην Επιτροπή μας. Ήθελα μόνο να επαναλάβω το εξής, ότι η ομάδα των οικολόγων πρασίνων αυτή τη θέση έχει υιοθετήσει να προωθήσει τον πρωταρχικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα καθοδηγήσει την αλλαγή στο διεθνές στερέωμα, να επαναλάβουμε τη δέσμευσή ε, του χρόνου και να ε, τονίσουμε ότι πρόκειται για μια πραγματική επένδυση για το μέλλον. Ευχαριστούμε. Ο Thank you, Ευχαριστώ. Γενικά συμφωνώ με όσα αναφέρθηκαν εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά. Μετά τα 20 χρόνια από το Ρίο βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση. Και στον τομέα αυτό συμφωνώ με την πρόταση των Πρασίνων γιατί νομίζω ότι αν ε, συναντηθούμε στη Βραζιλία που θα είναι η χώρα αμφιτρίωνας και εκεί γνωρίζουμε ότι αποψηλώνονται τα δάση και η Βραζιλία είναι τυπική περίπτωση, όχι μόνο η Βραζιλία, η Ινδονησία και άλλες χώρες, αλλά καθώς η Βραζιλία είναι η χώρα αμφιτρίωνας, θα μπορούσε να αποτελέσει το παράδειγμα και έτσι θα μπορούσαμε να δείξουμε ότι αν υπάρχει κάποια πολιτική συμφωνία μπορούμε να λάβουμε δράση για τα τροπικά δάση. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με τους πρασίνους. Δεν είμαι σίγουρος αν ε, πρέπει να είμαστε πιο κάθετοι και να πάμε πιο μακριά από την αρχική πρόταση ε, της δήλωσης, αλλά να είμαστε υπέρ σας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, ε, υπάρχει ένα τεχνικό προβληματάκι. Φαίνεται ότι χρειάζονται και τα μηχανήματα διακοπές. Τι να γίνει τώρα. Λοιπόν, τρία άτομα έχουν ζητήσει τον λόγο. τι είναι τώρα, όχι. Θέλατε να μιλήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ζητώ συγγνώμη και είμαι γρυπιασμένη. Ζητώ συγγνώμη για την βραχνιασμένη φωνή μου. Αλλεργία έχετε, έτσι, όχι γρήπη. Ναι, ναι, ναι, αλλεργία στη γύρι. Ε, η αποτελεσματική χρήση των πόρων, το πρασίνισμα της οικονομίας, αυτά είναι τα βασικά ζητήματα και πώς θα συνδυάσουμε την οικονομική διακυβέρνηση με την ε, αναπτυξιακή πολιτική. Εγώ δεν θα, ε, ε, Δεδομένε τη κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, δεν θα ασχολιόμουν τόσο πολύ με τη ΣΥΠΑ για το πρασίνισμα της οικονομίας ε, και θα καταθέσω και κάποιε κάποιες τροπολογίε. τροπολογίες. Πρέπει να είναι ισχυρότερο όπω η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των πόρων, κυρίως ω προς τους δείκτες και ως προς τη θέση των διαπραγματευτών μας σχετικά με την χρηματοδότηση στον τομέα του ε, περιβάλλοντος. Τελευταία παρατήρηση. Το θεματολόγιο των διαφόρων δράσεων που αναφέρατε θα μπορούσε ίσως να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει για μια ε, διεθνή συμφωνία για να έχουμε ε, εργαλεία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Πρόεδρος, παρακαλώ, έχετε ένα λεπτό έκαστος. Και μετά πρέπει να δούμε την έκθεση της κυρίας Οκονή για τον αθλητισμό, γιατί έχουν έρθει οι υπουργοί. Καμπριέλ Καμπράντε, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ πιέζομαι από το χρόνο. Λοιπόν, φαίνεται σαν να είναι μια επέτειος η διάσκεψη Ρίο στην 20, αλλά είναι πολύ καλή χρονική συγκυρία. Θέλω να τονίσω δύο πολύ σημαντικά θέματα αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα των πόρων. Καθημερινά στις εφημερίδες ε, γίνεται αναφορά για την έλλειψη των πόρων. Καθίσταται ένα τεράστιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην διάσκεψη Ρίο 20 να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, έτσι ώστε να αποφύγουμε να νηλοσκοτωθούμε για τους τρεις τελευταίους πόρους που θα υπάρχουν στο έδαφος. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την πράσινη οικονομία. Δεν ε, θεωρώ ότι η πράσινη οικονομία είναι κάποιο είδου υποοικονομία. Πρέπει να καταστήσουμε πιο οικολογική την οικονομία. Και νομίζω ότι αυτή η διάκριση είναι διαφορετική σε σχέση με αυτό που κλείνει πράσινη οικονομία. Τώρα για τι επιδοτήσεις. Ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταληξούμε σε κάποια συμπεράσματα από αυτού στη διάσκεψη του Ρίου ε, ξοδεύουμε 3 εκατομμύρια ευρώ για ε, επιδοτήσεις, επιζήμιες ε, και ακόμη περισσότερα για να εξαλείψουμε τα αρνητικά αποτελέσματα αυτών των επιδοτήσεων. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκέρεκ. Θα είμαι σύντομος. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φυσικά η συζήτηση αυτή και Πρέπει να πω ότι κάπως ε, όμως είναι απομακρυσμένη από την πραγματικότητα. Ζούμε σε μια οικονομία της αγοράς, υπάρχει ελεύθερο εμπόριο και υπάρχουν κάποιοι κανόνες που δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε. Η κυρία λύση για το πρόβλημα θα έγκυτω στο να αλλάξουμε το μοντέλο κατανάλωσης. Και δεν γίνεται και ιδιαίτερος λόγος γι' αυτό. το αμερικανικό μοντέλο είναι λανθασμένο και νομίζω ότι 20 χρόνια μετά το Ρίο πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε. Πρέπει να προωθήσουμε την χρήση των πράσινων τεχνολογιών κτλ. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι δυνατή αποτελεσματικότητα με τεχνολογία, αλλά η επάρκεια είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τροπολογίες μέχρι αύριο 12 η ώρα για να προλάβουμε να καταθέσουμε γέρο στην έκθεση. Θα ακούσουμε ακόμα την Σόφια Κονή για δύο λεπτά και η συζήτηση θα γίνει την άλλη φορά. Για να μην περιμένει ο κύριος Υπουργός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η συζήτηση για την έκθεση που συνδέεται με την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Αυτό είναι το θέμα. Όμω από την υπογραφή τη συνθήκη τη Λισαβόνα ξέρετε ότι συνιστά ευρωπαϊκή αρμοδία το αθλητισμό. Δεν ίσχυε αυτό μέχρι τούδε. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το στοιχείο, αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Ε, πρέπει να αναλυθεί από όλα τα μέλη τη επιτροπή μελλοντικά ούτω ώστε να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό ο αθλητισμός είναι εργαλείο στον τομέα της δημόσιας υγείας κυρίως ε, και πόσο σημαντικό είναι να καταπολεμήσουμε τη φαρμακοδιέγερση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό, όπως ε, έλεγα, ο αθλητισμός είναι ε, ένα βασικό θέμα προβληματισμού γενικότερα για την Ευρώπη. Περιμένω λοιπόν μια νέα συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσω την έκθεσή μου. Πριν το Στρασβούργο έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον Αύγουστο. Στο Στρασβούργο μου γνέφεται. Δεν γίνεται πριν το Στρασβούργο, Πρόεδρε. Ε, το περιμένω γιατί θα ήθελα να έχουμε μια επικοδομητική εκτεταμένη συζήτηση ή δυνατόν πριν το Στρασβούργο. Πρόεδρος, θα δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του αθλητισμού στην ε, κοινωνία μας. Ναι, μα ναι, γιατί είναι σημαντικό για την δημόσια υγεία. Είναι ένα εργαλείο αθλητισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει δημόσια συζήτηση. Ε, ευχαριστούμε και τώρα θα καλωσορίσουμε την, τον εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας. So, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τη χαρά να καλωσορίσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Νέα Πολωνική Προεδρία και τον ε, Υπουργό Περιβάλλοντος, ε, τον κύριο Αντρέη Κρασεύσκη. Καλώς στην Επιτροπή μας, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ και πολλά χρόνια ήταν κινητήριος δύναμη για μια καλή ποιότητα ζωής, για υψηλά πρότυπα κατά των ζημιογόνων εκπομπών. Καλωσορίζουμε λοιπόν την νέα Προεδρία και σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας όταν επισκέφθηκε την προσωπία μας στην Βαρσοβία. Έχουμε πάρα πολύ καλές αναμνήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι ο υπουργό είναι ταυτόχρονα και καθηγητή πανεπιστημίου στη Βαρσοβία και είχαμε και ένα δείπνο αργά τη νύχτα μέχρι τα μεσάνυχτα και βέβαια θα πάω τώρα στο σπίτι και 8 η ώρα το πρωί θα πάω στο Πανεπιστήμιο για να δώσω μαθήματα για την εφόρο ανάπτυξη. Και έτσι όπω μα είπε και χτε στην άτυπη υπουργική συνεδρίαση, ότι ε, μπορεί οι φοιτητέ να μην πηγαίνουν στα άλλα μαθήματα, αλλά στο μάθημά του είναι 100% η προσέλευση. Έτσι λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχει πραγματική δέσμευση ε, σχετικά με το συνολικό θέμα για το πώς θα πετύχουμε την αιφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας και στον κόσμο. Και ολοκληρώσαμε τώρα μόλις τη συζήτηση για τη διάσκεψη Ρίος 20 που θα λάβει χώρα από την Προεδρία της Δανίας ε, και βέβαια θα ε, ακούσουν και οι συνάδελφοι τι γίνεται στο τρίο της Προεδρίας, πώς συνεργάζεται με τη Δανία και την Κύπρο. Έτσι λοιπόν, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα έχει πολλά δύσκολα θέματα μπροστά τη Πολωνική Προεδρία. Έχουμε και την διάσκεψη των ημερών 17, την COP17 στην Νότια Αφρική, την προστασία του κλίματο. Έχουμε τον οδικό χάρτη για την αποδοτικότητα των πόρων το Σεπτέμβριο. Και θα έχουμε και τη στρατηγική τη βιοποικιλότητα. Μεγάλα ζητήματα λοιπόν επιτάπητο. που αφορούν ε, και την νομοθεσία, αλλά θα έχουμε και άλλα θέματα που θα προτείνετε εσείς κατά τη διάρκεια του ξαμήνου. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Σας δίνω το λόγο τώρα για την παρουσίασή σας. Thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Τζο. οι καθηγητές, ε, ξέρετε, θεωρούν ότι έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 45 λεπτά μονοκοπανιά, χωρίς να σταματήσουν. Οπότε δώστε, δώστε μου λίγο χρόνο. Αξιότιμοι βουλευτές. Εδώ εκπροσωπώ την Πολωνική Προεδρία, όπως γνωρίζετε, που θα προεδρεύει στο ε, ε, Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος ε, και Κλιματικών Αλλαγών για το επόμενο εξάμεινο. Επίσης, ανήκω στην κυβέρνηση μιας μεγάλης χώρας που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να αναπτυχθεί ταχύτατα σε όλους ε, τους τομείς. Πολιτιστικά, περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά, αναπτύχθηκε η χώρα μας ε, με γοργούς ρυθμούς. Και ε, Νιώθω ιδιαίτερο ενθουσιασμό που μπορώ να συμμετάσχω τώρα στις ε, εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτούς ε, τους τομείς. Εξάλλου έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία 60 ε, χρόνια στην Πολωνία. Όπως φαίνεται από διαδοχές δημοσκοπήσεις η κοινή γνώμη τάσεται σαφέστατα υπέρ της ευρωπαϊκή Ένωσης με την προσχώρησή μας μπορέσαμε να κάνουμε επενδύσεις ε, για τις ε, εθνικές μας υποδομές. Μπορέσαμε επίσης να εφαρμόσουμε την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία όπως εφαρμόζεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι στον τομέα των υποδομών ε, και του περιβάλλοντος έχει σημειωθεί πρόοδος αντίστοιχη με αυτή που κατέστησε δυνατή το σχέδιο Μάρσαλ ε, στο παρελθόν. Θεωρούμε πως με αυτήν την πολιτική ε, που θα ακολουθήσουμε στην Προεδρία θα αποπληρώσουμε το χρέος μας σε εισαγωγικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αν την ευκαιρία της Προεδρίας ε, λοιπόν για να ε, αποπληρώσουμε αυτό το ε, χρέος προς την Ένωση. Τα περιβαλλοντικά θέματα συνδέονται άρρηκτα με τα κοινωνικά και τα πολιτικά ζητήματα και ως εκ τούτου ε, δεν ε, μπορούμε να τα αναλύσουμε ξεχωριστά. Είναι αλληλένδετα όλα αυτά τα θέματα, οι κλιματικές αλλαγές και οι προκλήσεις ε, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινέ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Έχουμε ε, υπερβολικά μεγάλη εξάρτηση από την εξόρυξη άνθρακα. Η προστασία του περιβάλλοντος ως προς τις κλιματικές αλλαγές ε, είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Μας ικανοποιεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε σε αυτό το τομέα, διότι έχει ηγετικό ρόλο ε, στην ε, διεθνή σκηνή για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας εμείς ε, θα προαγάγουμε αυτό το ρόλο της Ένωσης. Ε, ταυτόχρονα υπάρχουν νέοι ανταγωνισμοί με τις ε, αναδυόμενες οικονομίες. Ε, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία αλλάζουν τα δεδομένα. Η παγκόσμια τάξη θα αλλάξει εντός ολίγου και οι κλιματικές αλλαγές ε, είναι ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την παγκόσμια οικονομία. Το κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να αναλυθεί όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και μακροοικονομικό πώς το θέμα της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος και το κόστος που αυτό συνεπάγεται έχει ιδιαίτερο ε, διότι αν δεν επομιστούμε εμείς το κόστος τότε θα μετακυλιστεί σε επόμενες γενιές με πολλαπλασιαστικό όμως αποτέλεσμα δυστυχώς. Εάν δεν πληρώσουμε το λογαριασμό εξάλλου, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα που παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα στις προσπάθειες αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Οι εκπομπές μας κυμαίνονται στο 12-13%. Θα χάσουμε τον αγώνα εναντίον ε, των οικονομικών δυνάμεων που πιστεύουμε ότι πρώτα πρέπει να τραφούν και μετά να καθαρίσουν. Σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να πιέσουμε για μια νέα δεσμευτική συμφωνία που θα προσυπογράψουν όλες οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές, ε, κυρίως η Κίνα και η ΙΠΑ που ε, έχουν το 50% των εκπομπών διεθνώς. Δεν πιστεύουμε ότι στην 17η Σύνοδο των Συμβαλωμένων Μερών στον Τέρμεν θα μπορέσουμε να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία. Παρόλα αυτά, τα κράτη-μέλη θα συνεργαστούν ούτω ώστε να υπάρξει σε πρώτη φάση μια προσέγγιση των εθνικών θέσεων, μια σύγκληση των εθνικών θέσεων. Μπορούμε να επιδιώξουμε να ε, παρατείνουμε την ισχύ του πρωτοκόλλου του Κιώτο Και επίσης θα ασχοληθούμε με το θέμα ε, της ε, χρηματοδότησης ε, και του Πρασίνου Ταμείου Green Fund ε, που συμφωνήθηκε στην Κανκούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, καλείται να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν θα διαβουλευτεί με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών που έχουν τις υψηλότερες εκπομπές θα πρέπει να διευκρινίσει ότι θα ακολουθήσει τη γραμμή της Ένωσης προσπαθώντας να ε, επιτύχει μια μείωση των εκπομπών. Και ε, σε αυτά τα πλαίσια το βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντεπεξέλθουμε είναι να δημιουργήσουμε νέα βιομηχανία που θα βασίζεται σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες. Η Κίνα και η Αμερική ήδη ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία και βραχυπρόθεσμα νομίζω ότι αυτό θα επιφέρει οικονομικά ωφέλη. Το δυναμικό ως προς τις επενδύσεις και την έρευνα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από κράτος σε κράτος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. πριν ε, αναλάβουμε φιλόδοξες δεσμεύσεις, επειδή έχουμε ηγετικό ρόλο, θα πρέπει να αναλύσουμε προσεκτικά το κόστος της περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο ένωσης και ανά ε, τομέα οικονομικής ε, δραστηριότητας που απειλείται από την διαφυγή, τη διαρροή του άνθρακα. Δεν θα έπρεπε οι ισχυρότερες οικονομίες να υποφεληθούν και οι ασθενέστερες να τα σπασμένα. Η πολιτική προστασία του περιβάλλοντος ε, και η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών δεν θα έπρεπε όμως να οδηγήσουν σε αύξηση της ανεργία σε άλλους κλάδους. Η Πολωνία δεν είναι κατά αυτής της πολιτικής, ε, αλλά ε, θα μελετήσουμε τα στατιστικά δεδομένα που θα μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα, διότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ε, οι ασθμένουσες ε, οικονομίες κάποιων χωρών αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης βλάπτουν, επηρεάζουν αρνητικά συνολικότερα την οικονομία της Ένωσης. Και η Πολωνική Προεδρία δεν πιστεύει ότι η αύξηση των πόντων ε, των δικαιωμάτων ε, των ε, εκπομπών μπορεί να μας οδηγήσει σε μείωση της δρύπανσης. Στις ασθενείς οικονομίες δεν υπάρχουν κονδύλια για επενδύσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι επενδύσεις στις καινοτόμες τεχνολογίες θα αποτύχανε αν εμείς διοχετεύσουμε όλα τα διαθέσιμα κονδύλια στην παραγωγή ενέργειας και στα δικαιώματα εκπομπών. Θα υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Ναι, σε αυτό το τομέα μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. και ε, οι επενδύσεις μας μπορούν να καρποφορήσουν ταχύτατα. Αυτό επηρεάζει την βαριά, την ελαφριά βιομηχανία, τα νοικοκυριά ε, και όλους τους υπολείπους ε, κλάδους πέραν της πληροφορικής. Ε, συγγνώμη, και όλους τους υπολείπους κλάδους πέραν του συστήματος εκπομπής ρήπων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικές. Ξέρω ότι αφιερώνω πολύ χρόνο στο θέμα τη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, αλλά είναι θελημένο γιατί είναι μέγιστε οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε πριν τον Τέρμπαν. Όμω και σε άλλου τομεί υπάρχουν βασικέ προκλήσει και άρα οι υπόλοιπε προτεραιότητε τη πολιτική Προεδρία είναι παραδείγματο χάρη η αποδοτική ε, χρήση των ε, ενεργειακών μα πόρων. Πρόκειται για βασική προτεραιότητα της Προεδρίας. Ε, παρατηρούμε μια κατασπατάληση των φυσικών πόρων λόγω του τωρινού ε, συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης. Ακολουθούμε μια ε, λανθασμένη ε, προσέγγιση, κατακαιρματισμένη προσέγγιση των πόρων. Ε, εξάγουμε δηλαδή ε, τους πόρους, επεξεργαζόμαστε, τους καταναλώνουμε και τους απορρίπτουμε. Κάποια κράτη-μέλη έχουν μεγάλη επιτυχία ε, κατά την προώθηση μιας οικονομίας που βασίζεται στον κύκλο ζωής ε, των προϊόντων. Ε, όμως θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρικότερη θεώρηση. Δείτε την εκθετική ανάπτυξη που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Είτε μιλάμε για το ΑΕΠ, είτε για την χρήση των πόρων η, ανάπτυξη, ε, η αναπτυξιακή πορεία επιταχύνεται κάθε χρόνο ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και αν δεν καταφέρουμε να βρούμε από τον Άρη πλουτόνιο ή αργό πετρέλαιο από την Αφροδίτη, θα χρειαστεί να ε, τα καταφέρουμε με τους πόρους που διαθέτουμε. Άρα θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις για δύσκολα ζητήματα όπως αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι εδώ έχει ηγετικό ρόλο και η Ένωση αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειδικότερα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξηγήσει πώς η ανάπτυξη ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο δείκτης ε, του ΑΕΠ ως μοναδικός δείκτης για την ε, καταμέτρηση της πρόοδου. Χρειαζόμαστε άλλους τρόπους παραγωγής προϊόντων που έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής, παραδείγματος χάρη. Είναι απαραίτητη η διαπαιδαγώγηση των νέων καταναλωτών, ενό νέου είδους καταναλωτών. Χρειαζόμαστε καταναλωτές που δεν θα θέλουν να αλλάζουν κινητό τηλέφωνο κάθε χρόνο, και ε, δεν θα ε, βγάζουν άχρηστο το πλυντήριο παραδείγματο χάρη μετά από τρία χρόνια. Ε, ένα, μια μεγάλη επιτυχία του Κοινοβουλίου ήταν ο οικουμενικός φορτιστής για τα κινητά τηλέφωνα. Άλλο πολύ σημαντικό θέμα, η βιοπικιλομορφία. Είναι ένα θέμα που συνδέεται με την βιώσιμη ανάπτυξη και φυσικά θα συζητηθεί στην ε, συνδιάσκεψη Ρίο συν Η Προεδρία μας θα συντονίσει τις κοινοτικές θέσεις. Έχουμε ένα εξάμεινο στη διάθεσή μας για να εκπονήσουμε μια κοινή θέση. Καλωσορίζω την ε, βούληση του ε, Κοινοβουλίου να παρουσιάσει τη θέση του και να την ε, προωθήσει κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της Πολωνικής Προεδρίας Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ήδη έχουμε ε, ξεκινήσει αυτό το δρόμο της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε στον τρόπο λειτουργίας μας. Στην Ευρώπη επιθυμούμε μια πράσινη οικονομία. Μάλιστα, στην ε, Πολωνία ε, θεωρούμε ότι μόνο μέσα από την πράσινη οικονομία θα απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Άρα κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η βιοπικιλότητα είναι ένας ε, τομέας όπου έχουμε σημειώσει πρόοδο κατονομάστε μία άλλη χώρα, ένα άλλο μέρος του κόσμου, όπου 20% της επικράτειας έχει το καθεστώς του Natura 2000, του προστατευόμενου βιότοπου δηλαδή. Χρειαζόμαστε περίπου πενταπλάσια κονδύλια στον προϋπολογισμό μας για να προστατεύσουμε αυτούς τους βιοτόπους και την ε, βιοπικιλότητα. Εν κατακλείδη. Έχω πλήρη επίγνωση το ότι θα θα συνεργαστούμε στενά για την εκπόνηση νέων νομοθετικών πράξεων. Εγώ θα είμαι ο πιστός και αφοσιωμένος υπηρέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο εξάμεινο και θα συνεργαστώ μαζί σας για θέματα όπως αναθεώρηση της οδηγίας για τα ηλεκτρονικά απόβλητα, Επίσης, αναθεώρηση του κανονισμού ΠΙΚ. Θα μπορούσα να σας μιλάω ένα 20 λεπτό για κάθε ένα από τα επιμέρους ε, ζητήματα, αλλά δεν θα το κάνω. Ήθελα μόνο να τονίσω η σημασία έχει συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να σημειωθεί τα στα πρόοδος. Πριν ε, αναλάβω το αξίωμα του Υπουργού Περιβάλλοντος, κατάφερα να ρυθμίσω διάφορα προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη μια παρακαμπτήρια οδός στην ε, βορειοανατολική Πολυνέα που θα περνούσε μια, μέσα από μια ελώδη περιοχή. και προσφέρω τις υπηρεσίες μου, ε, μπορώ να λειτουργήσω ως διαμεσολαβητής, ως διαπραγματευτής Είμαι στη διάθεσή σας. Προσφέρω τις υπηρεσίες μου για να γεννηθεί ο νέος κανονισμός που φυσικά θα είναι μεγάλη επιτυχία και της Πολωνικής Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. θα μιλήσω γερμανικά, βάλτε τα ακουστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και... Ακούσαμε πραγματικά τα μηνύματά σας, τα μεγάλα θέματα που απασχολούν και εμάς. Καλώς ορίζουμε ολόκληρη την ομάδα της Πολωνικής Προεδρίας. Αναφέρατε την αποτελεσματική χρήση των πόρων και το πλυντήριο του Υπουργού που έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Ευρώπη γιατί έχει ένα πλυντήριο πάνω από 30 χρόνια και εξακολουθεί να λειτουργεί έξοχα. Ένα παράδειγμα που αναφέρθηκε στη, στο Συμβούλιο Υπουργών για να υπάρχει κατανάλωση χωρίς πατάλη. Και να μην πετάμε τα πράγματα πριν χαλάσουν. Αναφέρατε την προστασία του κλίματος. και το ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεσολάβηση γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν ε, έχουν όλοι τις ίδιες ιδέες, την ίδια φιλοδοξία αλλά πρέπει να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια φωνή, το είπατε, δεν έχουμε ελπίδα εάν πάμε στον Τέρμπαν με διαφορετικές ε, φωνές. Το έχει δείξει αυτό και το παρελθόν. Πρέπει να έχουμε ένα μήνυμα ως Ευρώπη για ε, να διατηρήσουμε ηγετικό ρόλο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό και να προσπαθήσει ο καθένας γι' αυτό. Ε, βιοπικιλότητα, το ξανατονίσατε, ε, είπατε τι ωραίο τοπίο έχει η Πολωνία, όπου τα πράγματα είναι ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση και βλέπετε τι γίνεται με την δασοκομεία, τη γεωργία, την προστασία της φύσης, ένα μεγάλο θέμα βέβαια για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχουν πάρα πολλές καταστροφές και αλλαγές. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς ορίζω και τους συνεργάτες σας. Έχουμε λοιπόν μία σειρά Α, τώρα ερωτήσεων με τρία λεπτάκια λοιπόν. Πρώτα απ' όλα Πέτερ Λίζη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου για την εισαγωγή σας. Έχω κάποιες σύντομες ερωτήσεις για την προστασία του κλίματος. Σήμερα το πρωί εδώ πέρα έγινε μια μικρή συζήτηση. Ο πρόεδρος μας είπε πως ε, στο Συμβούλιο υπήρξε κριτική ή τουλάχιστον απορία για το ότι εμείς ως ε, Κοινοβούλιο δεν υιοθετήσαμε ψήφισμα τη βδομάδα που μας πέρασε. Απορώ κάπως και θα ήθελα να σας ρωτήσω ως πρόεδρο του Συμβουλίου, πώς αιτιολογείται την κριτική που ασκήθηκε στο Κοινοβούλιο, γιατί αν μας ενημερώνουν σωστά, το Συμβούλιο ότως ή άλλως και αυτό δεν μπόρεσε να συμφωνήσει και η δική σας κυβέρνηση έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Οπότε θα ήθελα μια διευκρίνηση από εσάς. Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο όσον αφορά τη μη συμφωνία του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, είπατε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν ρόλο ηγετικό στην προστασία του κλίματος. Ε, θέλω να τη αιτιολογήσετε αυτό γιατί πλέον δεν είναι τόσο πιστευτό. Έχουμε ένα στόχο 25%. Η Βραζιλία έχει ένα ρόλο 36 με 39% κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο περιμέναμε από τις χώρες αυτές το 2007 οπότε πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και όταν δεν είμαστε τόσο φιλόδοξοι όσο θεωρούμε. Τέλο πάντων, δούμε τώρα το μέλλον. Σωστά αναφερθήκατε στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Αυτό σχετίζεται άμεσα με τους στόχου του κλίματος. Τι προγραμματίζει συγκεκριμένα η πολεμική Προεδρία. Γιατί καλά τα είπε ο κύριο Σέτιγκερ ε, όλοι του πανηγυρικού μια χαρά τα λέμε, αλλά όταν φτάνει η ώρα των πράξεων στο Συμβούλιο Υπουργών, ε, είναι όλοι κατά. Τότε τι προγραμματίζει συγκεκριμένα η Πολωνική Προεδρία και μετά η σχέση μεταξύ στόχων αυτών και ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Είπατε σωστά και το υποστηρίζω πως πράγματι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα σε μεγάλο μέρος είναι εκτός του εμπορίου εκπομπών π.χ. στα κτίρια. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει κάποιο effort sharing σε αυτή την περίπτωση. Αν δηλαδή επιτύχουμε κάποιες πολλές ε, ε, οικονομίες, τότε δεν ε, μοιράζονται όλοι εξίσου το βάρος. Γιατί λέτε πως εμείς αναμφισβήτητα είμαστε ηγετική δύναμη, δεν ισχύει αυτό. Και Τέλος, ο Πέτερ Λάιος, ο οποίος εκπροσωπεί τώρα, ήταν συνάδελφός μας και εκπροσωπεί την Ουγγαρία στο Συμβούλιο, έκανε μια μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ουγγαρία και κατέληξε σε πολύ θετικό αποτέλεσμα. Τη γνωρίζετε αυτή τη μελέτη και υπάρχει κάτι ανάλογο για την Πολωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε πρώτα μερικές ερωτήσεις πριν να ακούσουμε απαντήσεις. Κοιτάξτε, δεν ήταν το Συμβούλιο να το ξεκαθαρίσω, όχι επισήμως ε, που άσκησε κριτική. Υπήρχαν διαφορετικοί διάφοροι υπουργοί, μάλλον οι οποίοι απόρρισαν για το ότι δεν επιτύχαμε συμφωνία. Δεν ήταν η επίσημη θέση του Συμβουλίου, αλλά υπήρχε μία διήμερη συνεδρίαση και απορούσε ο... απορούσαν μερικοί με το τι συνέβη. Λοιπόν. Εσείς κατόπιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό Περιβαλλόντος της Πολωνίας ε, και να ευχηθώ καλή τύχη στην Πολωνική Προεδρία. Θα ήθελα να αναφερθώ στο περιβαλλοντικό σχέδιο, το περιβαλλοντικό σχέδιο, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνδέει το περιβάλλον με τους βιώσιμους στόχους, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ε, και γνωρίζετε ότι υπάρχει και η περιβαλλοντική συνιστόσα για την κοινωτική στρατηγική για την έξυπνη ανάπτυξη. Και ξέρω ότι εσείς θα διδραματίσετε ένα σημαντικό ρόλο στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το επόμενο περιβαλλοντικό σχέδιο, το 7ο, γιατί το σημερινό θα λήξει στα τέλη του 2012 και θέλω να μου πείτε τι αναμένετε από την αξιολόγηση του ΕΚ του περιβαλλοντικού σχεδίου και ποια θα είναι η συνέχιση αυτήν την ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ σημαντική ερώτηση, κυρία Λεπάζ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για που παρευρίσκεστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την πρότασή σας να έχετε ένα ρόλο διαμεσολαβητή για τα κλιματικά ζητήματα, ξέρετε ότι ανησυχούμε κάπως να βλέπουμε μία μεταβαλλόμενη πολιτική βούληση και ε, για το ότι αυτός ο ηγετικό ρόλος για την Ευρώπη το κλίμα δεν είναι και απολύτως πραγματικότητα. Εγώ συμφωνώ εδώ με τον κύριο Λίζε τους επόμενους μήνες της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Ε, πώς ε, θα προχωρήσετε και πώς θα παντρέψετε ένα πολιτικό λόγο με την πραγματικότητα στην πράξη και ξέρετε πόσο σημασία δίνουμε στα θέματα τα ενεργειακά. Τώρα, για του ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια πριν κάποιες μέρες ψήφισε την ε, έκθεση που είχε θετήσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, κατόπιν δική μου πρόταση. Τώρα το μπαλάκι είναι στο κήπεδο του Συμβουλίου. Εσείς σκοπεύετε να ξανασυζητήσετε το θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας δηλαδή έτσι ώστε ο πρόεδρος Μπαρόζο και η Κομισιόν να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και νομίζω ότι κάποιοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Και τρίτο σχόλιο. Προετοιμασία της διάσκεψης Ρίο 20. Αναφέρθηκε και ο πρόεδρος Λάινεν στην εισαγωγή του στο θέμα αυτό. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να ε, φτάσει πέρα από τα ωραία λόγια σε κάποιες ε, προτάσεις συγκεκριμένες που θα συνοδεύονται και από την ε, κατάλληλη χρηματοδότηση ή πιστεύετε ότι θα παραμείνουμε σε αυτά τα ωραία λόγια. Κερδίσατε και χρόνο πρώτα. Δεν χρησιμοποίησα όλο το χρόνο στη διάθεσή μου. σα. ευχαριστώ λοιπόν για το λεπτό αυτό που μου ας ο κύριος Μύρος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Θέλω να αναφερθώ στην προετοιμασία της διάσκεψης ε, του Ντέρμπαν. Πριν δύο έτη, η Ευρωπαϊκή έθεσε το στόχο της ε, ενεργειακής αυτάρκειας για την Πολωνία και για τη χώρα μου. Η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο είναι μεγάλο πρόβλημα. Εμφανίστηκαν ορισμένες λύσεις, ανέκυψαν ορισμένες λύσεις οι οποίες παρόλα αυτά δεν είναι ικανοποιητικέ ε, από τη σκοπιά της περιβαλλοντικής προστασίας, όπως παραδείγματος χάρη αέριο όπως παραδείγματο χάρη. Ποια είναι η άποψή σας ε, για τα πολωνικά σχέδια στον τομέα αυτό Ποια είναι η άποψή σα για τη χρήση τη πυρηνική ενέργεια για την καταπολέμηση τη ε, κλιματική αλλαγή, κυρίω ε, για την κατάσταση στην Ευρώπη, κατόπιν ε, τη απόφαση Γερμανία να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ, Σάτου Χάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό που προσήλθε για να συζητήσουμε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Καλή επιτυχία για την Προεδρία σας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ε, δεν είναι πολύ ενθαρρυντική η αρχή. Είπατε, Υπουργέ, πως ε, θέλετε να συνεχίσει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας η Ένωση να έχει αυτό τον ηγετικό ρόλο. Αλλά όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ο κύριος ε, και η κυρία Λεπάζ, Ο ρόλος ε, της Πολωνίας ε, τις περασμένες εβδομάδες στο Συμβούλιο δεν ήταν ιδιαίτερα ε, θετικός από αυτή τη σκοπιά στις δηλώσεις σας δε άκουσα κάποια σταθερά πάγια επιχειρήματα της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων. Ξέρετε, θα τεθεί σε κίνδυνο η ίδια η λειτουργία της κοινωνίας αν υπερβούμε τους δύο βαθμούς Κελσίου. Στην Κανκούν δεν επαρκούν αυτές οι δεσμεύσεις των κρατών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να αυξήσουμε ε, τα όρια όπως θα συμφωνηθούν στην Κανκούν για τις εκπομπές. Ε, αν ε, λέτε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε ως πρότυπο αυξάνοντας τις δεσμεύσεις μας, τότε ποια είναι η στρατηγική σας λοιπόν για να το υλοποιήσετε, πώς ε, θα περιορίσετε τη μείωση σε κάτω από δύο βαθμούς Κελσίου την αύξηση συγγνώμη, της θερμοκρασίας σε κάτω από κελσίου ή μήπως βαθμούς Κελσίου ή μήπως θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντική η βιομηχανία των ορεικτών καυσίμων σε σχέση με τα ε, σημερινά παιδιά της Πολωνίας, ε, τα εγγόνια σας ας πούμε. Ε, πρόεδρος, ε, ακούσατε πέντε ομιλητές από πέντε διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Αν θέλετε, απαντήστε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε άλλους δέκα που Θέλω να σας θέσουν ερωτήσεις. Μην μακρηγορήσετε για να προλάβουμε να τους ακούσουμε όλους. Παρακαλώ. I will try to be very... Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν, να αναφερθώ στο θέμα του 25%. αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί όχι στην Προεδρία, αλλά από το λαό θα ήθελα να σας καθησυχάσω. ότι δεν είναι η πρόθεσή μας ε, να υπερασπίσουμε εδώ τα συμφέροντα των ε, λόμπι ε, για τα ορχεία στην Πολωνία. Τα λόμπι αυτά δεν είναι πλέον τόσο ισχυρά όσο στο παρελθόν. τα λόμπι της εξορρυκτικής βιομηχανίας δηλαδή. Εμείς ε, κατανοούμε ότι είναι αναπόφευκτη μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ξέρουμε ότι πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το λιγνίτη. Και ακόμη και πριν από την δημοσίευση του δικού χάρτη για το 2050, γνωρίζαμε ότι το 40% του λιγνίτη ήταν ε, το μέγιστο το οποίο θα μπορούσε να θέσει οικονομία μας. Τώρα πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτή τη στρατηγική. Και θέλω να εξηγήσω γιατί θέσαμε βέτο στο σχέδιο του 25% από την Κομισιόν, γιατί δεν ε, είχαμε τα απαραίτητα στοιχεία, τις απαραίτητες μελέτες και αναλύσεις. σε σχέση με τον οικονομικό αντίκτυπο στα μη μονομένα κράτη-μέλη. Ζήτησα τα στοιχεία αυτά πέρσι τον Ιούνιο και μου υποσχέθηκαν ότι μια ανάλυση αναχώρα θα δημοσιευόταν, θα υλοποιούταν, αλλά ποτέ τελικά δεν μας έδωσαν αυτά τα δεδομένα. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην Κοπενχάγη συμφώνησαν ότι υπό ορισμένε ε, προϋποθέσεις θα ήταν ε, υπέρ μεγαλύτερων στόχων μείωσης θέλω να πω στους κυρίους Χέση και Λίζε ότι εμείς κάναμε πάρα πολύ προσεκτικά τους υπολογισμούς μας σε ό,τι αφορά ε, το πόσο θα κοστίσει στην πολεμική οικονομία ο στόχος του 20%. Είναι μεταξύ του 1,9 και 1% του ΕΠ. Ε, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες τη Παγκοσμία Τράπεζα έκαναν του ίδιου υπολογισμού και κατέληξαν ε, σε πιο απεσιόδοξα αποτελέσματα μεταξύ του 1,2 και του 1,4%. Τώρα, αν ε, ρωτήσω συναδέλφου από άλλες χώρες αν έχουν τέτοιους υπολογισμούς, απαντούν αρνητικά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μέχρι να μάθουμε ποιες είναι οι συνέπειες των αποφασεών μας δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιλέξουμε μια κατάσταση η οποία θα επιδεινώσει σημαντικά την οικονομία μας. Και δεν μιλώ μόνο για τον άνθρακα. Αν ε, πρέπει παραδείγματο χάρη να καταβάλουμε επιδόματα ανεργία ε, σε ένα μεγαλύτερο αριθμό, αριθμό ανέργων, αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τομέα του άνθρακα. Τώρα για το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή είναι η πρώτη μας επιλογή. Προς εκεί πρέπει να κατευθυνθεί η Ευρώπη καταρχήν. Και θα πρέπει η προσέγγιση να είναι ευρεία. Πιστεύω ότι η εμπειρία της Πολωνίας θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα σε άλλες χώρες. περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται ΥΟΣ από το Ταμείο Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Πολωνία για θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις επιχειρήσεις ε, έχουν χρηματοδότηση 40% για ηλιακά πάνελ, παραδείγματο χάρη. Εμείς ε, προσφέρουμε ευφυή e, πράσινη ανάπτυξη και επίσης χρηματοδοτούμε πολλά άλλα προγράμματα, όπως ε, προγράμματα για τη μόνωση των κτηρίων. Όποιο κτίριο χρήζει μόνωσης είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Τώρα, κύριε πλούμ για το έκτο περιβαλλοντικό πρόγραμμα, ναι, θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό η Προεδρία το επόμενο εξάμεινο. Θα πρέπει να εκπονήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση για την αξιολόγηση του έκτου προγράμματος την άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, το ΣΟΠΟΤ, ε, συζητήθηκε το θέμα αυτό και ακούστηκαν και κάποιες επικρίσεις. Δόθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι δεν πετύχαμε. Όμως, παρόλα αυτά δεν υπήρχε ούτε μία φωνή, και το γνωρίζει αυτό ο κ. Λάινεν, ούτε μία φωνή δεν υπήρχε από κάποιον από τους 27 υπουργούς ή επικεφαλής αντιπροσωπιών κατά του 7ου προγράμματος. Δηλαδή, ακόμη και αν το 6ο πρόγραμμα δεν ήταν απόλυτα επιτυχές, ίσως ακόμη και αυτό να αποτελεί ένα καλό λόγο για να έχουμε το 7ο πρόγραμμα. Ίσως θα πρέπει να καταβάλουμε διπλές προσπάθειες και να, παρέχουμε, να παράσχουμε περισσότερους πόρους για να διασφαλίσουμε ότι την επόμενη φορά θα πετύχουμε όσο δεν πετύχαμε αυτή τη φορά. Φυσικά, το 7ο πρόγραμμα θα υφετηθεί από την Προεδρία της Δανίας, ε, η οποία θα αναλάβει τη σκητάλη της Προεδρίας από εμά. Τώρα, κοινή θέση πριν τον Τέρμπαν. Τι ήθελα να αναφέρω Κάτι που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπω ε, ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν ε, επισκέπτεστε ε, άλλα κοινοβούλια για να πείστε τους συναδέλφους να δράσουν από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση για συντονισμένη δράση και συντονισμένες φιλοδοξίες, προς ε, πολιτικά δεσμευτικές συμφωνίες. Νομίζω ότι αυτό είναι ο δικός σας σημαντικός ρόλος και μπορείτε να βοηθήσετε πάρα πολύ όταν τα κοινοβούλια διάφορων χωρών ε, και κυρίως ε, όσων εκπέμπουν περισσότερο να συνενωθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αισθανόμαστε κάπως εγκατελειμμένοι για διάφορους λόγους. Κάθε χώρα, η Πακίνα, η Ιαπωνία, και κάθε χώρα έχει διαφορετικά επιχειρήματα γιατί δεν μπορούν να συμβαδίσουν μαζί μας, γιατί γιατί πρέπει να είναι πιο πίσω από μας. Έτσι λοιπόν αυτός είναι ο μεγάλος ρόλος που έχει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, να προχωρήσω στην ώρα της κυρίας Λεπάζ. Εδώ θα μπορούσα να διαδραματίσω ένα ρόλο μεσολαβητή. Είμαι πάρα πολύ καλός ε, στο να καταλήγω σε λύσεις μέσω διαπραγμάτευσης. Και πάντοτε προσπαθώ να σφυριλατήσω ένα συμβιβασμό στην Πολωνία ως υπουργός περιβάλλοντος. Κατόρθωσα να διαμορφώσω την νομοθεσία μας για τους γάμματα αφομικρών με έναν τέτοιο τρόπο που μας επέτρεψε τον πειραματισμό. Εγώ είμαι επιστήμονας, πιστεύω στα πειράματα και στη μάθηση δεν υπάρχει λόγος να απαγορεύσουμε τις εισαγωγές γαματαφόμικρων, μικρών, το χάρη μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών, αλλά δεν είμαι υπέρ του να απελευθερώσουμε τους γαματάφ όμικρον στο περιβάλλον. Δεν μπορούμε να παραβιάσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υπό την πολωνική νομοθεσία δεν είναι δυνατό να έχουμε ούτε, ένα τετραγωνικό καλλιέργεια γαματάφα ομικρών και νομίζω ότι αν στην Πολωνία προχωρήσουν τα πράγματα θα είναι πιο εύκολη η κατάσταση. Τώρα, Ρίο 20. Θα μπορέσει η Ευρώπη να κάνει περισσότερα πέρα από το να εξτομίσει ωραία λόγια. Ευχαριστώ κυρία Λεπάζ για την ερώτησή σας γιατί και εγώ έχω αμφιβολία σχετικά. Δεν ξέρω αν ε, είμαστε έτοιμοι για το νοητικό άλμα. Είμαστε τόσο συνηθισμένοι να ανανεώνουμε κάθε χρόνο το κινητό μας. Ε, πραγματικά μας ε, συναρπάζει κάθε νέο μοντέλο αυτοκινήτου που βγαίνει στην αγορά. Καταρχήν πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό μας. Και νομίζω ότι θα συμφωνούσατε μαζί μου. Αλλά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Δεν θα μείνουμε στα λόγια. Έχουμε συμφωνήσει σε συγκεκριμένε δράσεις. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε και αποτελέσματα. Θα πρέπει τις δράσεις μας να τις καταστήσουμε πραγματικότητα. Σε σχέση με το αέριο σχιστόληθο. Η ερώτηση του κυρίου Όσκα. Κοιτάξτε, το base load ναι, ναι, ναι, energetics είναι κάτι αναμφισβήτητο. δηλαδή ενέργεια με βασικό φορτίο. Δηλαδή είναι κάτι που μπορούμε να δημιουργήσουμε και με τα φωτοβολταϊκά. Ε, Συγγνώμη, η βασική ενέργεια που πρέπει να παρέχει το δίκτυο είναι κάτι αναμφισβήτητο. Έχουμε και τι ανανεώσιμε πηγέ ε, ενέργεια, αλλά πολλέ φορέ μπορεί να μην φυσήξει ο άνεμο. Ε, τώρα έχουμε και το λιγνίτι και άλλες μορφές ενέργειας, ε, αλλά παραδείγματο χάρη σε κάποιες χώρες της Ευρώπης δεν είναι της μόδας. Ε, στη Βόρεια Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, δεν μιλάμε για το λιγνίδι, υπάρχει πυρηνική ενέργεια. Όμως με τη Φουκουσίμα κανείς δεν τη θέλει την πυρηνική ενέργεια. Και έχουμε και το συμβατικό φυσικό αέριο. Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την εξαρτησή μα στο ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά δεν το κάνουμε αυτό στην Πολωνία και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρώπη οθέτησε την άποψη ότι δεν θέλει να εξαρτάται 100% από το ρωσικό αέριο. Αν δεν ε, μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να υποφεληθούμε από το αέριο όπως και στο όλυθο, θα πρέπει τελικά να χρησιμοποιούμε κεριά για να διαβάζουμε τη νύχτα. Η αλήθεια είναι ότι και οι τέσσερι πηγέ ενέργεια έχουν τα προβλήματά τους, έχουν μειονεκτήματα και πρέπει να τα αξιολογήσουμε αυτά τα μειονεκτήματα. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ιδανική πηγή τέτοιας βασικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ενεργειακό μείγμα αναχώρα που θα μας δώσει επαρκή ενέργεια, ανταγωνιστική και θα μπορούμε παράλληλα και να προστατεύουμε το περιβάλλον. Σας διαβεβαιώ ότι έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες, έχουμε ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα στην Πολωνία για τις περιβαλλοντικές μελέτες αντικτύπου και κάποιοι λένε ότι μάλιστα και πολύ αυστηρό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, είναι ρομαντικό να διαβάζει κανείς με το κερί, αλλά δεν είναι πολύ πρακτικό. Ελπίζουμε τις επόμενες ε, δεκαετίες, οι επόμενες ε, πηγές ενέργειας, ήλιος, αέρας, βιομάζα, βιοθερμία, γεωθερμία, να μπορέσουν με τις κατάλληλες πηγές, με τις κατάλληλες τα αποθηκευτικά μέσα να μας παρέχουν ενέργεια. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τις επόμενες ερωτήσεις, δύο λεπτά maximum. Λοιπόν, Καρλ Χάιντς Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε του Συμβουλίου, να σας συγχαρώ. Είστε ο 25ος πρόεδρος του Συμβουλίου που συναντώ και μετά την παρουσίασή σας ανήκετε πραγματικά στις ε, εντυπωσιακέ περιπτώσεις. Ε, λοιπόν, Ποιο είναι το πιο σημαντικό σας χάρτης ε, για το Ντέρμπαν, όχι το Κανκούν, συγγνώμη, ναι, το, το Κανκούν με, με ακόμα. Τι λέτε στους ε, ομολογούς σας ε, στο Συμβούλιο Υπουργών και τι συνιστάτε στην Επιτροπή μας. Ε, όπως ε, λέτε, θέμε όλοι να μιλήσουμε με μία φωνή. Δεύτερον, εγώ είμαι ο κακός με τα ηλεκτρικά απόβλητα. Εγώ κληρονόμησα τον πλητήριο από τη μάνα μου. η μεγαλύτερη συσκευή που υπάρχει εκεί πέρα στο, στο αγρόκτημα. Οπότε να σας πω επίσης πως ε, να συγχαρώ για το ότι ο συνεργάτης σας ήρθε 8 η ώρα στο πρωινό για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, Βεβαίω. θα να μάθω και ποια είναι η θέση σας ε, για τη σχέση και με τις υπόλοιπε ε, χώρε. Εντάξει, δεν συμφωνείτε οπωσδήποτε με το Κοινοβούλιο, αλλά δεν συμφωνείτε και μεταξύ σα όλοι στο Συμβούλιο. Εκεί πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Καρλ Χαντσλόντσε. Ευτυχώ που τελικά είχε ένα ραντεβού με την ε, Πολωνική Προεδρία. Λοιπόν, Κρήτον Αρσένη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας καλωσορίσω, Υπουργέ. Ε, είστε υπέρ της Ευρώπης ε, στην Πολωνία και σας καλωσορίζουμε στην ε, Προεδρία. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει να βρούμε κοινέ λύσεις για τα κοινά μας προβλήματα. Όπως και οι συνάδελφοι για τις κλιματικές αλλαγές θα συμφωνήσω και θα πω ότι πρέπει να ανταγωνιστούμε πρώτα απ' όλα ε, με χώρες που ασχολούνται με το να τραφούν πρώτα πριν λύσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και αναφερθήκατε κυρίως στην Κίνα. Ναι, αλλά η Κίνα έχει ριζοσπαστικά μέτρα. Κλείνει εργοστάσια που, χρησιμοποιούν τεχνολογία που εμείς ακόμη χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή. Κλείνουν τα εργοστάσια στην Κίνα όμως. Σήμερα δεν νιώθουμε ίσως απελημένοι από τον ανταγωνισμό της Κίνας, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Ποιος θα ανταγωνιστεί την πράσινη Κίνα του αύριο, αν ε, χάσουμε αυτόν τον αγώνα. Γιατί με την ε, αξία της αγοράς ε, μιλάμε για 13. Αυτό είναι το κόστος. Ε, για την πολιτική ε, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Μπορεί να μην συμφωνούμε με την προσέγγιση της Κίνας, αλλά εκείνοι κάτι κάνουν. Εμείς τι κάνουμε. Αν δεν βρούμε λύση, χάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας, την ανάπτυξή μας, τις θέσεις απασχόλησης. Καταλαβαίνω γιατί τονίζεται ιδιαιτέρως ε, πόσο σημαντικό είναι να μειώσουμε την κατανάλωσή μας. Ναι, συμφωνώ, αλλά με αυτούς τους στόχους μείωση θα κατοχυρώσουμε και τη μείωση της κατανάλωσης. Θέλω να συμφωνήσω και με την ερώτηση του κυρίου Φλόρενς. Με ποιο τρόπο ακριβώς ε, προτίθεστε να επιτύχετε την ε, μείωση της κατανάλωσης, τη μείωση των εκπομπών και την ομοθυμία ενόψη του Ντέρμπαν ε, για τα τέλη του έτους. Σας ευχαριστούμε. Κύριος Κεμπάντη. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, Υπουργέ Κρασέσκη. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που επέκριναν, κατέκριναν τη θέση σας ε, για τις ε, κλιματικές αλλαγές. Εγώ έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο χάνουμε την ηθική, από ηθικής πλευράς ηγετική θέση που έχουμε, αλλά θα υποφέρουμε και οικονομικός πώς αν δεν δράσουμε σύντομα. Σε λίγα χρόνια θα πρέπει να αγοράζουμε τεχνολογία από την Κίνα, από την Ιαπωνία και άλλες χώρες που θα έχουν προχωρήσει πολύ σε σχέση με την Ευρώπη. Είμαι εισηγητής για το θέμα της αποδοτικής χρήσης των πόρων και πολύ θα ήθελα να συζητήσω αυτό το θέμα μαζί σας, αλλά καλύτερα να περιμένουμε τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν αρχίσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κάτι για ένα άλλο προσφύλλες για μένα ζήτημα, βιοπικιλομορφία, βιοπικιλότητα. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο ε, λόγω της τάσης του Συμβουλίου. Ε, πέρσι στην Αγκόγια ε, είχαμε τους, ε, ήταν απρόσμενα καλά τα αποτελέσματα, θέσαμε τους στόχους και στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος όμως κρατημέλη δεν ήθελαν να συζητήσουν αυτούς τους στόχους. Η Ολλανδία, η χώρα μου, συζητούσε για στόχους για τους οποίους έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια κτλ. Ναι, ναι, βεβαίως η χώρα που κάνει, πετυχαίνει μία μείωση 60% στον προϋπολογισμό της, καταλαβαίνετε δεν έχει πολλά διαθέσιμα κονδύλια, οπότε το να είναι προσιτός ο στόχος δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Εσείς μιλήσατε για ένα κόστος που θα αυξηθεί στο μέλλον αν δεν δράσουμε τώρα βεβαίως και στον τομέα της βιοπικιλότητας αυτό αληθεύει όλους ιδιαίτερος και σας ε, ρωτώ το εξής, τι θα κάνετε ούτως ώστε το Συμβούλιο όχι μόνο να εγκρίνει τους στόχους αλλά και να τους ε, εφαρμόσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά του και να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη όπως πριν από μια δεκαετία. Σας ευχαριστώ, ε, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σόνικ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να, επιστρέ... να επανέλθω σε ένα ζήτημα που ανέφερε ο υπουργό. Οι περιοχές Natura 2000 ε, συχνά είναι ιδιωτικές εκτάσεις. Και οι ιδιοκτήτες συχνά θεωρούν ε, την περιοχή Natura 2000 ως μπελά. που δεν τους επιτρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Ήδη στην προηγούμενη θητεία μιλάμε για την ανάγκη περισσότερων πόρων για να προστατεύσουμε τις περιοχές ε, Natura 2000. Βλέπετε λοιπόν όρεξη στο Συμβούλιο για να αυξηθεί αυτή η χρηματοδότηση. Ευχαριστώ Ματίας Γκρότε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις δηλώσεις σας. Άκουσα προσεκτικά του κοινωνικού κόστους ε, της ενέργειας και της κλιματικής πολιτικής. Κοιτάξτε, ε, έχω αντιληφθεί σωστά, συμφωνείτε μαζί μας πως θα πρέπει για όλα αυτά τα πράγματα να υπάρχουν μελέτες κοινωνικών επιπτώσεων από την Κομισιόν. Ε, θα είστε στο πλευρό μας. Το ερώτημά μου τώρα, Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία. Πολλοί ε, συνάδελφοι τοποθετήθηκαν, αλλά μήπως θα έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερη κλιματική διπλωματία η Ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα στον Τέρμπαν. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να έχουμε κάτι με τους ε, παγκόσμιους εταίρους μας, όχι κάτι μετά το Κιώτο, να προσπαθήσουμε για μια συμφωνία η οποία θα είναι πραγματικότητα. Η κλιματική πολιτική συνολικά και στην Ευρώπη έχω ορισμένε φορές την εντύπωση πως δεν έχει τα απαραίτητα μέσα και δυνατότητες ανάλυσης. Παραδείγματο χάρη, όταν οι επιχειρήσει πραγματικά θέλουν να πουν το, και να ανακαλύψουν το πραγματικό αποτύπωμα των προϊόντων ε, δεν υπάρχουν ε, μέσα. Θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο για να δούμε τι θα γίνει ε, με απτά μέσα για να υπάρχει μια συγκρισιμότητα και των προϊόντων και να ξέρει και το κοινό ότι υπάρχει στο χύψη προϊόν σε αυτό το μπουκάλι από πλευράς διοξιδίου του άνθρακα και μπορεί να γίνει νομίζω και εξαγωγική επιτυχία εάν είμαστε εμείς οι πρώτοι. Και σας παρακαλώ να είστε πιο ε, φιλόδοξοι και όσον αφορά την κλιματική πολιτική και να κάνουμε ένα βήμα προ τα εμπρός. Ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω πως οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Δευτέρα στη συνεδρίασή τους ε, συζήτησαν το θέμα του κλίματος Οπότε η εξωτερική πολιτική νομίζω απασχολεί την εξωτερική πολιτική να απασχολεί αυτό το θέμα. Λοιπόν, Ρίτα Μάνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ για την εξαιρετική αυτή κίνηση και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τις εκπομπές ε, των πλοίων ε, και την οδηγία σχετικά με τις ε, εκπομπές των οξυδίων του θείου. Υπάρχει μια απόφαση από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας ε, να μειωθούν αυτές οι κομπές θείου από τα πλοία. Φυσικά κάτι τέτοιο το καλωσορίζουμε, αλλά υπάρχει μια σειρά προκλήσεων για το μέλλον ε, της ναυτιλίας των θαλάσσιων μεταφερών. Μία από τις αδυναμίες ε, της απόφασης του ΕΜΟ είναι ότι ε, αντιμετωπίζει διαφορετικά τις διάφορες περιφέρειες, τις διάφορες περιοχές. Θα το γνωρίζετε φαντάζομαι. Μέχρι το 2015 αυτές οι εκπομπές του θείου θα πρέπει να μειωθούν σε ορισμένες ε, περιοχές Σε ορισμένε περιοχέ πρέπει να μειωθούν 0,1 ενώ σε άλλε περιοχέ 0,5. Οι στόχοι. Ο στόχο μα είναι να έχουμε του ίδιου στόχου για τι μειώσει παντού, σε όλο τον κόσμο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Υπουργό, ποια είναι η άποψη τη προεδρία για αυτή την οδηγία για τις ε, εκπομπές εξωτερικού του θείου και πόσο ενεργά ασχολείται η Προεδρία με το θέμα αυτό θέμα για την Βαλτική. Ξέρετε, έχουν ληφθεί αποφάσεις και αντιδρά κάπως η ναυτιλία. Λοιπόν, Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του. Είναι πάρα πολύ σημαντική κυρίως έχοντας ε, κατά νου τον Τέρμπαν, ε, πραγματικά μας βελπίζει έτσι λοιπόν ε, πραγματικά βασιζόμαστε στις ε, ικανότητές σας να μεσολαβήσετε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι πρέπει να πάμε στον Τερμπέν με μια απάντηση στη δήλωση του Μπαλί, δηλαδή ε, να έχουμε κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τώρα δεν ε, έχει υπάρξει μία πρόταση που να βασίζεται στην κλιματική δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, εγώ σας ζητώ να αντιμετωπίσετε και να αναλάβετε την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η μόνη δυνατότητα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το Κιώτο. Αν ε, θέλετε θα μιλήσουμε λεπτομερέστερα σε άλλες περιπτώσεις ε, για το συμπέρασμα, δηλαδή ένα άτομο, ένα δωρεάν δικαίωμα εκπομπών. Αυτή είναι η απάντηση και εγώ θεωρώ ότι αυτή η απάντηση πρέπει να δοθεί στη δήλωση του Μπαλή. Από την άλλη, πιστεύω ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξετάσουμε τον οδικό χάρτη για μια Ευρώπη χωρίς ε, άνθρακα μέχρι το 2050. Αν ε, είναι αλήθεια αυτό, αν μπορούμε να προχωρήσουμε από μόνοι μας, τότε αυτό αλλάζει το κοιότο. γιατί εγώ πιστεύω ότι τότε θα μπορούσαμε να πούμε ας προχωρήσουμε για δικό μας λογαριασμό και μπορούμε και να αλλάξουμε εντελώ τη θέση μας και να πούμε αν ε, οι άλλοι δεν ε, συμμετέχουν, ας ε, πάμε στον αλλακτικό σχέδιο, δηλαδή να έχουμε ένα ποσοστό, μάλλον να περιοριστούμε εμείς και να έχουμε και ένα φόρο σε ό,τι αφορά τον άνθρακα. Εγώ έχω θέσει αυτό το ερώτημα σε πάρα πολλά άτομα μέχρι τώρα. Δεν έχω λάβει μέχρι τώρα απάντηση. Ελπίζω από εσά να τη λάβω. Ο κύριο Υπουργό ήταν και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, οπότε ξέρει Ιταλικά. Φρανσό Γκροστέλ. Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Μας ε, είπατε προηγουμένως ε, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον άνθρακα για να έχουμε κάποια ε, ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά θα έπρεπε να περιορίσουμε ε, τη χρήση του άνθρακα. Φυσικά δεν ε, δείχνεται αυτό αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, αλλά έχουμε μία μέθοδο, έχουμε νέες τεχνολογίες με την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε αυτό το πρόβλημα του άνθρακα και δι του αερίου, του φυσικού αερίου. Ξέρουμε ότι έχετε διάφορα σχέδια. Ε, έχουμε όμως αυτές τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες, ε, λειτουργούν αισίως, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε και να βρούμε τη χρηματοδότηση, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει οικονομική δέσμευση. Από πολιτική σκοπιά ε, υπόσχεστε να ασκήσετε τη μέγιστη δυνατή πίεση ώστε να βρεθεί η χρηματοδότηση, να βρεθούν τα κονδύλια και να χρησιμοποιηθεί αυτή η νέα τεχνολογία στην Ευρώπη και να έχουμε και το τεχνολογικό προβάδισμα σε σχέση με την Κίνα και τη ΣΥΠΑ, γιατί και αυτές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Μισελ Ριβαζή, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Υπουργέ, που ήρθατε για να απαντήσετε στι ερωτήσει μα. Πριν από ένα δεκαπενθήμερο πήγα στην Πολωνία, ακριβώ για να αξιολογήσουμε την ενεργειακή πολιτική. Και ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό το φυσικό αέριο ισχύ Εφόσον είσαστε η, ναυαρχίδα, αν θέλετε, στον τομέα αυτό, γιατί έχετε εκδώσει 90 άδειε για την εκμετάλλευση φυσικού αερίου από σχιστόλιθο ήδη, είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε τι γίνεται με, τις, ε, ε, με τα υπόγεια ύδατα και τους υδροφόρους ορίζοντες. Ε, πώς, ρωτώ, θα ενισχύσετε την προστασία των υπογείων υδάτων μετά την εξόρυξη. Δεν μιλώ καν για την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Δηλαδή χρησιμοποιούνται 500 έως 600 χημικά προϊόντα, ε, νευροτοξικά, έτσι, τοξικά κτλ και κατόπιν ε, τα πόνερα με κάποιο τρόπο θα πρέπει να τα χειριστούμε και προς το παρόν δεν υπάρχουν ε, μονάδες καθαρισμού λιμάτων. Πώς γίνεται να έχουμε ε, ε, κανόνες ε, για τα οξύδια του αζότου, παραδείγματος χάρη, να μην έχουμε όμως κανένα κανόνα για αυτά τα χημικά προϊόντα. Άλλη ερώτηση. Μας μιλήσατε για το ρωσικό αέριο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αλλά με το αέριο σχιστόλιθο θα εξαρτάστε από τη ΣΥΠΑ, γιατί εκείνοι έχουν το δίπλωμα εύρεση τεχνίας για την κατασκευή των μονάδων. και σε επίπεδο Πολωνίας ε, Πώ ε, θέλετε να ακολουθήσετε αυτή την οδό ενώ ουσιαστικά θα αυξηθούν οι εκπομπέ. Τώρα τελευταίο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. είναι γιατί δεν είδα ούτε ε, φωτοβολταϊκά, δεν είδα ούτε ανεμογεννήτριες στην Πολωνία. Είδα μια μεγάλη μονάδα βιομάζας. Εντάξει, αλλά χρειάζεται και εσεί ενεργειακή διαφοροποίηση. Αφού μα μιλάτε για ενεργειακό μίξε, μείγμα, ας αναπτύξετε λοιπόν τι απαιτούμενε τεχνολογίε τεχνολογίε για να επαναβιομηχανοποιήσετε κλάδου που έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία για την Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίρικ έχει ζητήσει επίση το λόγο πριν να ακούσουμε τον Υπουργό. Μινίστα, αλλά ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό, κυρίως υπό την ιδιότητα του καθηγητή η Πολωνική Προεδρία αποτελεί ευκαιρία να ακουστούν καλύτερα οι μορφωμένοι άνθρωποι. Δυστυχώς, πολλές φορές η Ευρώπη κοφεύει, ακούει μόνο τις ομάδες των λόμπι. Το διακυβερνητικό πάνελ της IPCC για την κλιματική αλλαγή παρουσίασε μια υπόθεση που η Πολωνική Ακαδημία Επιστημών απέριψε. Η IPCC ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη μόνο μία μεταβλητή του διοξιδίου του άνθρακα, ενώ υπάρχουν ε, πάρα πολλές μεταβλητές. Το δόγμα της ε, IPCC Ήδη έχει επιπτώσει στη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη ε, καθημερινή ζωή. Υπάρχει ένα φάντασμα ε, των εκπομπών διεξουδίου του άνθρακα. Αυτή είναι η επίσημη ιδεολογία. Ήρθε η στιγμή να υπάρχει ένα επιστημονικό πάνελ για κλιματικά ζητήματα. Θέλω να ρωτήσω, είναι δυνατόν. καθώς ε, προετοιμαζόμαστε για τη Βραζιλία και εν ώψη του Ντέρμπαν πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάσκεψη, πρέπει να προστατεύσουμε το κλίμα αλλά και τους πολίτες. Μάλιστα ακούσαμε όλο το φάσμα των απόψεων που υπάρχουν στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή ε, από επιστήμονα σε επιστήμονα. Θα προσπαθήσει τώρα να απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Σε 15 λεπτάκια γιατί μετά πρέπει να ολοκληρώσουμε. Szanowni ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλόρενς για τις ε, προσπάθειες που κάνει σχετικά με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρονικών ε, συσκευών, ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών. και ο κλάδος, ε, η βιομηχανία συνεργάστηκε μαζί μας ε, για να ε, δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων. Η οδηγία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Φλώνης καθότι ήταν και ο εισηγητής. στην αναθεωρημένη εκδοχή της θα αντισταθμίσει, θα καλύψει τις ατέλειες του της πρώτης οδηγίας. Ως προς τις φιλοδοξίες που έχουμε εν ώψη της διάσκεψης του Ντερμπέρνα και τη διατήρηση αυτής της ηγετική θέσης από πλευράς της Ένωσης, ε, θα σας έλεγα το εξής αξιότιμοι βουλευτές. Εάν η Κίνα υλοποιήσει τα σχέδιά της, δεν θα απολέσουμε το τον ηγετικό ρόλο γιατί θα έχουμε σημειώσει επιτυχία ε, στον τομέα της προστασίας ε, του περιβάλλοντος κατά των κλιματικών αλλαγών. Ε, το αντίθετο θα ήταν καταστροφικό. Τώρα αν μιμηθεί την Ιαπωνική αναπτυξιακή πορεία η Κίνα, γιατί έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, δεν μιλάμε για 400 ppm, αλλά για πάνω από 1.500 ppm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο πλανήτης δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Δεν μπορεί να απορροφήσει τέτοιες εκπομπές. Σε συζητήσεις ε, που είχα στην ε, Κίνα αναφέραμε ότι ένα πενταετές ε, πρόγραμμα δράσης δεν είναι κάτι το εξαιρετικό ένα τέτοιο πενταετές πρόγραμμα δεν ε, αποτελεί σε καμία περίπτωση αντιστάθμισμα για την παραδοσιακή προσέγγιση δηλαδή να ανοίγουμε ένα εργοστάσιο που λειτουργεί με άνθρακα κάθε εβδομάδα. Επίσης, ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ μέλεται να μειωθεί από το 12% στο 7% και είπαν οι Κινέζοι ότι μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές, δηλαδή ε, επιβραδύνοντας την ανάπτυξή τους. όχι μόνο ε, ελοχεύει κίνδυνος να χάσουμε αυτήν την ηγετική αυτό τον ηγετικό ρόλο που έχουμε, αλλά ο κίνδυνος, ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος, είναι να ακολουθήσουν άλλοι το παράδειγμα αυτό. Το έγγραφο που διαπραγματευόμαστε δεν είναι ικανοποιητικό. Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για τον Τέρμπαν, συντονίζοντα τις 27 εθνικές θέσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να αποφασίσουμε πρώτα απ' όλα αν επιθυμούμε να προβλεφθεί μια, δε, μια παράταση της ισχύω του κιότο. Ε, Κιώτο. Αυτό ζητούν πολλοί εταίροι μας, ε, η Κίνα τουλάχιστον αυτό επιθυμεί. Η ομάδα G77 εξάλλου και η Κίνα αυτό ζητούν. Ε, η ΕΠΑ πάλι αποστασιοποιούνται τελείως. Αν παραμείνουν έτσι τα δεδομένα είναι κρίσιμος ο ρόλος της Ένωσης, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Τη Δευτέρα το συζητήσαμε αυτό το θέμα. και η άποψη που επικράτει προς το παρόν είναι η εξής. Εάν ε, προχωρήσουμε μόνοι μας, εάν πληρώσουμε μόνοι μας ε, το λογαριασμό, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί ε, παράταση της ισχύως του πρωτοκόλλου. Άλλοι πάλι ανησυχούν ότι δεν κάνουμε αρκετά στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η Κίνα ε, το επόμενο εξάμεινο ούτε η ΕΠΑ ούτε η Βραζιλία θα αναλάβουν αυτόν τον ηγετικό ρόλο το επόμενο εξάμεινο. Εμείς θα τον διατηρήσουμε η Ένωση, δηλαδή και τα 27 μέλη της. Θα ε, καταδείξουμε την προσήλωσή μας για την επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά όχι ε, μόνοι μας, γιατί το μόνο που θα καταφέρουμε είναι ε, να συνεχίζουν να ανοίγουν νέα εργοστάσια κάθε εβδομάδα. Αυτό ε, θα ήθελα να το πω ως απάντηση προς την ερώτηση του κυρίου Αρσένη. Για την ε, βιοπικιλότητα τώρα, την ερώτηση του κυρίου Γκεπράντη, εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη η αξία ε, των οικοσυστημάτων στο έκτο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δεν είχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα για τα οικοσυστήματα. Ένα υγιές οικοσύστημα είναι αυτό που επιθυμούμε. Γιατί αν δεν είναι υγιές το οικοσύστημα, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε εκατομμύρια για να διορθώσουμε την κατάσταση. Αυτό να πούμε στους υπουργούς όταν μας λένε ότι δεν έχουν κονδύλια για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Πρέπει να τους πείσουμε πως Σε αυτό έγινε η αξία ε, του οικοσυστήματος. Γλιτώνουμε έτσι δις, τρεις ευρώ μελλοντικά. Βλέποντας τα στατιστικά δεδομένα, ε, ορισμένες φορές την να τα αμφισβητήσω, αλλά όμως αληθεύουν το εξακρίβωσα. Είναι πρέπει να τονίσουμε πόσα θα χάσουμε αν δεν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Αν τους πείσουμε τους υπουργούς για την εξοικονόμηση χρημάτων, μόνο τότε θα βρούμε τα διαθέσιμα κονδύλια. Δεν είμαστε σε θέση τώρα να υπολογίζουμε την αξία ενός δάσους ή του καθαρού νερού. Στη, στην Ηνωμένα έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη δε, υπολογίστηκε το ποσό που εξοικονομούμε, τα δισεκατομμύρια που εξοικονομούμε ε, για την προστασία από τις ε, πλημμύρες, εάν ε, εγκαίρως φροντίσουμε τα, τους μικρούς ποταμούς, τα, τα Συνεχίζοντας, για τις άμεσες πληρωμές τώρα θα έλεγα ε, ότι έχουμε δώσει επιπρόσθετες άμεσες πληρωμές για τη διαχείριση ε, χώρων που προστατεύονται βάσει του Natura 2000. Επίσης ε, επιχορηγούνται οι γεωργοί που ακολουθούν τις ορθές αγροπεριβαλλοντικές πρακτικές και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και ο κανόνας. Πολύ. θεωρούν ότι είναι ένα βάρος ε, ε, τα ιδιότοποι που προστατεύονται από το Natura 2000. Ε, εγώ, ξέρετε, έχω το εξοχικό μου σε περιοχή Natura 2000, μα πρόκειται για ευλογία. Γιατί ξέρω ότι παραθερίζω σε ένα μέρος όπου δεν θα χτιστούν τα διπλανά λιβάδια. Τι ωραία που είναι, ξυπνάω το πρωί ε, και έχω την ηρεμία μου. Δεν έχω όμως τη δυνατότητα να πηγαίνω συχνά. Ε, εάν ε, δώσουμε τα σωστά κίνητρα στους γεωργούς θα αγωνιστούν μαζί μας. Είναι οι θεματοφύλακες της φύσης, εξορισμού οι γεωργοί. για τους ε, πρασίνους τώρα την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Μα τα λέω εγώ στους φοιτητέ μου αυτά και θα προσφέρω κατά τη διάρκεια της ε, Πολωνικής ε, Προεδρίας. Αν θέλετε, διαλέξει να σας εξηγήσω ότι μιλάμε για τη φύση συνολικότερα. Αλλά υπάρχουν δύο περιβάλλοντα, το φυσικό και το κοινωνικό. Ε, μιλήσατε για την παρακαμπτήρια αυτή οδό με, στην ελότ περιοχή της Πολωνίας. Ε, ξέρετε, όταν ε, ε, φτιάχνετε μία νέα υποδομή που συνδέει δύο ε, κοινότητες, δύο οικισμούς, θα πρέπει να λάβετε υπόψη το ότι αν γίνουν επενδύσεις θα επηγιστούν και άλλες ε, περιοχές ε, στην Πολωνία. Κάναμε αξιολόγηση αντικτύπου, φτιάξαμε νέες, ε, νέους δρόμους. αλλά δεν αλυσοδένονται ε, οι, οι λύκοι και τα πουλιά, ξέρετε, έξω από το Υπουργείο. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται γι' αυτό. πέρα από το φυσικό περιβάλλον υπάρχει και το οικονομικό περιβάλλον. Τι εννοώ, ωραία όλα αυτά τα ευχολόγια, αλλά πρέπει και να τα πληρώσουμε, να υπολογίσουμε το κόστος των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, ε, πολυκριτηριακή ανάλυση ε, ονομάζεται αυτό. Ανάλυση που βασίζεται σε ε, πολλά διαφορετικά κριτήρια. Δεν προσπαθούμε να βάλουμε ετικέτα με την τιμή πάνω στα πουλιά, δεν είναι αυτό, ούτε ε, πάνω σε έναν άνθρωπο που πεθαίνει ε, λόγω αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. Ποια μεθοδολογία ε, χρησιμοποιούμε. Μια μεθοδολογία που μας επιτρέπει να κάνουμε αντιπαραβολή του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος ελαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές διαστάσεις. Δηλαδή, γιατί φτιάχνουμε τον αυτοκινητόδρομο για να οδηγούν οι άνθρωποι και να το χρησιμοποιούν πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος του να μην φτιαχτεί ο αυτοκινητόδρομος. Εκπομπές, σε μείωση των εκπομπών τώρα του διοξιδίου του θείου. Ερικα Μάνα. Μέχρι το 99 ε, μέχρι το 89 μάλλον ε, ήταν τέτοιο το, τόσο πολιταρχικό το καθεστώς στην Πολωνία που δεν λειτουργούσε τίποτα. Έκτοτε όμως έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στον τομέα της μείωσης των εκπομπών των διοξιδίων του θείου και του αζότου. Είναι κάτι, ένας τομέας όπου έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, ε, δηλαδή το δικαίωμα ε, τα δικαιώματα εκπομπής ρήπων και το, το μηχανισμό εμπορία τους. Όσοι υπερβαίνουν τα όρια, όσοι υπερβαίνουν τα δικαιώματα που τους έχουν χορηγηθεί, ε, συνεισφέρουν σε ένα ε, ταμείο το οποίο ε, ανταμείβει όσους κατάφεραν να μειώσουν τις εκπομπές ρήπων. Βιτόριο Πρόντι. ευχαρίστως ε, να συναντηθούμε κύριε Πρόεδρε και να σας εξηγήσω ότι προτίθεται να κάνει η και Προεδρία για να καταστήσει τον Τέρμπαν ε, επιτυχία παγκοσμίως, μια επιτυχία για τον κόσμο. Θα είναι μια επιτυχία για τον κόσμο, για ολόκληρο τον κόσμο, αν είναι επιτυχία για την Ευρώπη. Ευχαρίστως ε, να σας εξηγήσω πώς θα το πετύχουμε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τον οδικό χάρτη για το 2050, και τη φορολογία για το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν νομίζω ότι είναι αδύνατον. Πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία για να μειώσουμε το αποτύπωμα του άνθρακα. Δεν είναι αδύνατο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πείσουμε και τον υπάλληλο κόσμο. Έχουμε το δικαίωμα στην Ευρώπη να λέμε ότι αν κάποιος έχει μετακατασταθεί από την Ευρώπη για να παραγάγει γυαλί κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη και μολύνει όσο θέλει, γιατί στην άλλη χώρα στην άλλη περιοχή δεν υπάρχει όριο ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τότε εμείς έχουμε δικαίωμα να επιβάλλουμε οικονομικές κυρώσεις ε, σε αυτόν τον ε, κατασκευαστή μέσω δασμών στα σύνορα. Εγώ χρησιμοποίησα στο διαδίκτυο ένα τέτοιο, μια τέτοια μέθοδο υπολογισμού για το αποτύπωμα του άνθρακα. Και έβαλα τη δική μου περίπτωση, παραδείγματο χάρη, ε, εγώ στο εξοχικό μου προσπαθώ να χρησιμοποιώ δυνατόν πιο οικολογικές μεθόδους για τη θέρμανση, όμως, δηλαδή και οξύλα, αλλά τελικά ήμουν εχθρικός απέναντι στο περιβάλλον, γιατί παρήγαγα πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν, όταν είδα τι έπρεπε να εγκαταλείψω, ήταν πολλά αυτά τα οποία, συνειδητοποίησα ότι είναι πολλά αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα. Δεν έχω τώρα χρόνο να φερθώ σε αυτές τις λεπτομέρειες. Αλλά Τέλο. πάντων, σας τα λέω όλα αυτά για να σα πω ότι αν ε, θέλουμε στην Ευρώπη να έχουμε χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα, θα απαιτηθούν πολλέ θυσίε παντού. Και τώρα, εν συντομία, για το αεροποσχιστόλιθο. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξαρτηθούμε από τις ΗΠΑ. Νομίζω ότι ένα είναι η εξάρτηση από ορισμένα διπλώματα βρεσιτεχνίας, αλλά η εξάρτηση από ένα μεμονωμένο προμηθευτή που μπορεί να ανοίξει και να κλείσει την κάνουλα όποτε θέλει αυτός, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εντελώς διαφορετική εξάρτηση. Δεν υπάρχει ιδανικός ε, τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο που να βλάπτει όσο δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. αναφερθήκατε και στον υδροφορορίζοντα, στα υπόγεια Στην ε, μόλυνση του υδροφορορίζοντα. Αλλά παραδείγματος χάρη υπάρχουν και κίνδυνοι ε, όταν ε, χτίζουμε επίσης ε, ένα πυρηνικό εργοστάσιο Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Ναι, φυσικά είμαι υπέρ των ελληνικών πάρκων, αλλά μέχρι να μάθουμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια αυτή. Μέχρι να μπορέσουμε να αποθηκεύουμε κιλοβατόρες σε βάτ, τότε, μέχρι τότε χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τις βασικές πηγές ενέργειας. Έτσι λοιπόν μπορεί να ζηλεύουμε τους είδους ε, για το 40% της ε, ενέργειας ε, της υδροηλεκτρικής. Αλλά δεν μπορούμε όλοι να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα, Κύριε Γκέρεξ, ό,τι αφορά το σκεπτικισμό, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι σκεπτικιστής απέναντι στο κλίμα, Καθηγητή είμαι. Έχω πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τη θεωρία ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και αν ε, είχα μια αποδείξη να δείξω ότι χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο έπεσαν θύματα συλλογικής, συλλογική συλλογικής ε, φαντασίωσης ή είχαν συμφωνήσει να κοροϊδέψουν όλο τον κόσμο αν είχαν τέτοιε ε, αποδείξεις τότε μάλλον και βαρύνοι του πετρελαίου του Τέξας ε, θα με πλήρωναν για να δημοσιεύσω τις αποδείξεις αυτές. Όμως υπάρχει πραγματικά φαίνεται με σαφήνεια ότι έχουμε ανθρωπογενείς αιτίε ε, για τις κλιματικές αλλαγές και φυσικά θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες αποδείξεις όσο περνάει ο καιρός. Είναι ε, χρονοβόρα η εκδήλωση της κλιματικής αλλαγής. Ε, Κατανονικά χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια για να εκδηλωθεί και εμείς παρατηρήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι, Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Νομίζω τελευταία μια μισή ώρα είχαμε μία πλούσια γενική συζήτηση διαφόρων συστημάτων που θέλουμε να λύσουμε και να προωθήσουμε. Μπορώ να σα πω πως το Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί για να είναι επικοδομητικό και επικοδομητικός εταίρος για την Πολωνική Προεδρία, οπότε σας εύχομαι κάθε επιτυχία και εύχομαι να τα ξαναπούμε στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο και ίσως και στην Επιτροπή ε, τη δική μας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ την ομάδα σας. Καλή επιτυχία στην Πολωνική Προεδρία.